Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρωινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Το πρώτο σημείο της πρωινής ημερήσιας διάταξη είναι η ενημέρωση για την αποστολή που πραγματοποίησε η Επιτροπή μας στην Ουκρανία πέρυσι 5 7 Δεκεμβρίου. Μια ενιαμελής αντιπροσωπή από την Επιτροπή μας επισκέφθηκε το Κίεβο στις αρχές Δεκεμβρίου και συνάντησε τον Ουκρανό Πρωθυπουργό μέλη της Ουκρανικής Βουλής, ε, υψηλούς αξιωματούχους της νέας Ουκρανικής ε, Διοίκησης, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ στην Ουκρανία στην καινούργια κοινοβουλευτική θητεία την ένατη, κάτι που δείχνει τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία, καθώς και στη συνεργασία της με την Ουκρανική Βουλή, τη Βέρχοβνα Ράντα. Η αποστολή μας μάλιστα ήταν και πολύ επίκαιρη, ε, εν ώψη της απονομής του βραβείου Ζαχάροφ στον Όλεξ Σέντσοφ ε, που είχε προηγηθεί μια εβδομάδα πριν την αποστολή μας και την ε, υψηλή διάσκεψη που θα γίνει στο Παρίσι με βάση τη διαδικασία της Νορμανδίας την επόμενη εβδομάδα. Από τα πιο αξιοσημείωτα σημεία της επίσκεψης ήταν η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, τον Ολέξη Χοντσάροφ, που επανεπιβεβαίωσε την προθυμία της χώρας του να συνεχίσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και τις μεταρρυθμίσεις γενικώ σε πολλούς κλάδους. Και στις συναντήσεις που είχαμε με τους κοινοβουλευτικούς ε, ομολόγους μας και εκπροσώπους της κυβέρνησης, ε, ε, επιβεβαιώθηκε ότι οι νέε κρανικέ αρχές θέλουν να συνεχίσουν τι μεταρρυθμίσεις των προκατόχων τους με φιλόδοξους στόχους σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνία σύνδεση και την ευάθυνση τη ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, εκφράσαμε την πλήρη μας υποστήριξη στην πορεία της Ουκρανίας και ε, επισημάναμε ότι αυτή η διαδικασία τούρμπο πολύ εσπευσμένης έγκρισης ε, νομοσχεδίων δεν θα πρέπει να περιορίσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τις διαβουλεύσεις με άλλους εμπλεκομένους, κυρίως ε, κοινωνία των πολιτών και think tanks και δεν θα πρέπει αυτή η εσπευσμένη διαδικασία να επηρεάσει την ποιότητα της νομοθεσίας άλλο ξεσημείο το θέμα ήταν η συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας ε, και θέμα η κατάσταση ασφάλειας. Επιβεβαίωσε την ισχυρή πολιτική βούληση του Προέδρου να, να τεθεί ένα τέρμα στην διαμάχη στην Ανατολή, στη σύγκρουση στην Ανατολή, όχι όμως πάση θυσία και σίγουρα όχι βάσει των ε, προϋποθέσεων που υπαγορεύει η Ρωσία. Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ επίσης εγκομιάστηκε ιδιαίτερως και διατρανώθηκε η προθυμία της Ουκρανίας να επιδιώξει τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Ε, βέβαια, ανάλογα με κάποια εσωτερικά σημεία της οργάνωσης και θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά κάποιων μελών. Επίσης, ε, ακούσαμε την έκκληση για ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στον Εύξηνο Πόντο. Οι Ουκρανοί εξέφρασαν ε, την ε, εκτίμηση τους ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανάγκη να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία προκειμένου να ενισχυθούν οι μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και εκτιμά ιδιαίτερα την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας και επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει τη συνέχιση της επιβολής των κυρώσεων στο καθεστώς της Ρωσίας. Διαπιστώσαμε λοιπόν προθυμία των ε, Ουκρανικών αρχών ε, για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ένα φιλοευρωπαϊκό πνεύμα και πορεία της Ουκρανίας και ενθάρρυνση της συνεργασίας ε, της διακοινοβουλευτικής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Βέρχοβνα ΡΑΔΑ. Επίσης, εγώ με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας θα σας ενημερώσω για την δέκατη συνάντηση που είχε η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ε, με ομολόγους μας από τη Βέρχοφνα Ράδα στο Στρασβούργο 18 και 19 Δεκεμβρίου του 2019. Δηλαδή λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ουκρανία. Ήταν πολύ επίκαιρη αυτή η συνάντηση γιατί συνεχίστηκε το πνεύμα των συζητήσεων που είχαμε στο Κίεβο και ήταν μια πολύ καλή συνεδρίαση με πολύ ευχάριστο πνεύμα και έθεσε ένα πολύ θετικό τόνο για το μελλοντικό μας έργο σε πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας. Αυτές λοιπόν ήταν οι ενημερώσεις από τις δύο από συνεδριάσεις και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μισελ Γκάλερ που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας στην έκθεση για την Ουκρανία. Κύριε Γκάλερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να τονίσω κι εγώ αυτό που είπατε στην ανακεφαλαίωση ως μόνιμος εισηγητής. Έχω επικεντρωθεί στην υλοποίηση του DCFDA, δηλαδή της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης για τις ελεύθερες συναλλαγές και σημαντικό ήταν να δούμε την στάση και την ε, κινητοποίηση της σχετικά νέας κυβέρνησης. Και γενικώ είμαι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αφιβολίες ότι και αυτή η νέα κυβέρνηση που αποτελείται κυρίως από ένα νέο κόμμα και κατά 80% από νέους βουλευτές, την έχει μια έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Πρέπει τώρα να δούμε πώς θα προχωρήσουν με την υλοποίηση. Ήδη έχουμε αναφέρει ότι οι κοινοβουλευτικές σύνοδοι και οι προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν σε ταχύτητα τούρμπο, δηλαδή σχετικά γρήγορα να γίνουν πρώτα τα πιο εύκολα, εκεί που υπάρχει στήριξη, πολιτική στήριξη για να προχωρήσουν σε αλλαγές και μετά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μειωθεί η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων. Το Είδαμε και στις εκλογές στην Ουκρανία, τονίστηκε σε όλους ότι θα πρέπει να αναλάβουν όλοι υπεύθυνα το ρόλο τους ως βουλευτές. Και σχολαστικά να φροντίσουν να εξετάζουν όλες τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Θα πρέπει η πολιτική βούληση δηλαδή να αντικατοπτριστεί και σε πράξεις απτές. Έχουν συμβεί βέβαια κάποια πράγματα που δεν ήθελε κανείς. Ένα παράδειγμα ήταν μάλλον, <clears throat> ένα παράδειγμα ήταν η κατάργηση κάποιων ε, νόμων από το σοβιετικό καθεστώς και κάποιοι νόμοι από την εποχή του Κρουστόφ. που όριζε διαφορετικά τα εγκλήματα και τον ποινικό κώδικα σε σχέση με την Ουκρανία. Δεν είχαν λοιπόν ε, ε, ακυρωθεί αυτά, δεν είχαν ανασταλεί, παρόλο που οι Ρώσοι είχαν πει ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει διάλογος για τα θέματα αυτά. Και εμείς στην πλευρά από την πλευρά μας στη Ραχοχναράντα έπρεπε να επιμείνουμε. ώστε να πάρουν πολύ σοβαρά εκεί και να αντιληφθούν οι Ουκρανοί το ρόλο τους ως βουλευτές. Ναι, μου κάνετε νόημα ότι πρέπει να κλείσω κάπου εδώ, θα το, θα το πράξω. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Απλώς ήθελα να σας ε, λοιπόν να ολοκληρώσετε, να περάσετε στο διατάφτα. Σήμερα έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε κάπως αυστηροί στο χρόνο αγόρευσης. Θέλει κανείς παρακαλώ το λόγο? Δεν βλέπω κανένα. Α. Oui, en tant que... Euh, Μάλιστα. Ως μέλος αυτής της αντιπροσωπείας και συμμετέχουν στην αποστολή, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις και να προσθέσω ε, κάτι στην εξαιρετική ενημέρωση που μας έκαναν οι δύο προλαλήσαντες. Πρώτον, ε, στη νέα διοίκηση και η νέα κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο ε, εντυπωσιαστήκαμε από μια μεγάλη διαφορά για μας, για τους Γάλλους δηλαδή. Έχουμε μια κυβέρνηση κυρίως τεχνοκρατών που απαρτίζεται από προσωπικότητες που διαπνέονται από την πεποίθηση ότι με ευφυΐα και ταχύτητα μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε ριζικά μια χώρα. Και αυτό πραγματικά ήταν συναρπαστικό για μας γιατί όντως υπάρχει ταχύτητα, όντως υπάρχει μια διορατικότητα και ταυτόχρονα ένας τεράστιος κίνδυνος που ελοχεύει και που είναι να αποκοπεί αυτή η κυβέρνηση τεχνοκρατών από την δημόσια, από την κοινή γνώμη, από το κοινό που δεν θα καταλάβει ίσως αυτές τις μεταρρυθμίσεις και θα αποξενωθεί. Και έτσι θα προσκρούσουμε στο παραδοσιακό ρήγμα ελίτ και λαού που μπορεί να είναι τεχνητό, αλλά δυστυχώς μερικές φορές ε, ασκεί πολύ αρνητική επίδραση στον πολιτικό βίο. Δεύτερο εντυπωσιακό σημείο που το επισημάνατε κι εσείς είναι η τη βούληση αυτού του επιτελείου αυτής της νέας κυβέρνησης ε, να καταλήξει σε συμβαστική λύση με τη Ρωσία. Και αυτό θα είναι θεμελιώδη σημασία για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτή η βούληση δηλαδή είναι δηλωμένη των Ουκρανών να τεθεί ένα τέρμα στην διαδικασία. Και αυτό θα είναι η κυλιδία αλήθως για την Ρωσική Ομοσπονδία και για τον Πούτιν. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλος κανείς να ζητά το λόγο, οπότε να ολοκληρώσουμε με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο επόμενο. Προηγουμένως όμως, να σας θυμίσω ότι η κυρίως πόρτα της αίθουσας δίπλα στο Προεδρείο θα παραμένει κλειστή ε, για να παραμένουν συγκεντρωμένοι οι ομιλητές μας. Μέχρι να ολοκληρωθεί λοιπόν η συζήτηση με του προσκεκλημένου ομιλητές, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τις πόρτες στα πλάγια για την είσοδο στην αίθουσα. Τεχνική διευθέτηση αυτή για να είμαστε απερίσπαστοι στην ακρόασή μας και να μην ακούμε το θόρυβο από τις πόρτες που βροντοκοπάνε. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης η θεώρηση για την εξέλιξη της πολιτικής ε, ανατολικής γειτονίας μετά το 2020. Έχουμε μια δημόσια ακρόαση για την ανατολική γειτονία και τις ε, προβλεπόμενες εξελίξεις μετά το 2020. Ας περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα για να μπορέσουν να μπουν οι ομιλητές και να καθίσουν στο Προεδρείο. Um, Ευχαριστώ. Επαναρχόμαστε στο θέμα μας. Το 2019 ήταν η δέκατη επέτειος της Ανατολικής Γειτονίας. Ήταν όμως και μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, όπως φάνηκε από τις ευρεία, ευρείας και κάποιες φορές απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις, την ε, δυσφορία και την ανησυχία στα πολιτικά πράγματα και τι εκλογέ που μεταμόρφωσαν τι χώρε αυτέ. Το 2020 πιστεύουμε ότι επίση θα έχει πολλέ προκλήσει για πολλέ χώρε με ε, τοπικέ και κοινοβουλευτικέ, αλλά και προεδρικέ εκλογέ από τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το σημαντικότερο γεγονό θα είναι η σύνοδο για το μέλλον τη Ανατολική Γειτονία που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες την Άνοιξη. Εν ώψη λοιπόν αυτή τη Συνόδου, όπω είχαμε κάνει και το 2017, το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει έκθεση με συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εισηγητή τον κύριο Αστρεβίτσιους. Η ακρόαση λοιπόν αυτή είναι ε, άκρος επικαιρή. Επιτρέπει να μελετήσουμε μαζί τα επιτεύγματα και τις ελλείψεις της Ανατολικής Γειτονίας 10 χρόνια μετά την έναρξή της, αλλά το πλέον σημαντικό να αποτιμήσουμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα και καλύτερα για να υποστηρίξει τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας στις θεμητές ευρωπαϊκές τους βλέψεις. Προτού δώσω το λόγο στον εισηγητή για μια σύντομη εισήγηση, θα ήθελα να καλωσορίσω τους τέσσερις προσκεκλημένους ομιλητές μας για σήμερα. Τον κύριο Σέργη Γκερασίμτσουκ, που είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου για τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές σπουδές ε, στο Ουκρανικό πρίσμα, ε, τον κύριο Κορνέλη Κακάσια, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών ε, στο Πανεπιστήμιο του, της Τυφλίδας Ιβάνε στη Γεωργία, την κυρία Σινικού Κασάρη, η οποία είναι πολιτική αναλήτρια στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τις ε, Σπουδές Ασφάλειας, τον κύριο Κλάδιος Μανιώκας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου της συμβουλευτικής εταιρείας ESCP, Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Νομικά και Οικονομικά Προγράμματα, καθώς και ε, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους. Επίσης, για να εμπλουτίσουμε αυτές τις παρουσιάσεις, έχουμε προσκαλέσει και την κυρία Ματέρνοβα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Διεύθυνσης για την Κοινωνία και την Διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα... καθώς και την κυρία Αντζελίνα η οποία είναι διευθυντής ε, της υπηρεσίας για την ε, Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και τις σχέσεις με τη Δυτική Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία στην ΕΕΔ. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Έχετε πέντε λεπτά για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας, κυρία Στρεβίτης. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Γειτονία είναι ένας εμοχλός σταθερότητας και ειρήνης συχνά μας απασχολεί η επιτυχία και η προοπτική της. Οι χώρες της ανατολικής Τερικής σχέσης, της ανατολικής γειτονίας δηλαδή, ε, βρίσκονται σε μια ζώνη άμεσης ευρωπαϊκής ε, ε, επιρροής και αντιμετωπίζουν ένα φάσμα εξευρωπαϊσμού. Τα πρώτα βήματα, παρότι ήταν αργά και λιγότερο παραγωγικά, έχουν επιταχυνθεί και έχουν σημαντικό γεωπολιτικό αντίκτυπο στι ε, χώρε με τι οποίε έχουμε διαπραγματευτεί συμφωνίε σύνδεση με ολοκληρωμένε διευθετήσει ε, ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, ιδίω μετά το 2014. Η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία έχουν γίνει ενεργοί εταίροι και έχουν περάσει από εκβάθρων ε, οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις με διαφορετικά βέβαια αποτελέσματα ανάλογα με την εποχή. Η συνεργασία με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν γίνεται περισσότερο κατά περίπτωση με συμφωνίες επιμερισμένων συμφερόντων, με στενούς οικονομικούς δεσμούς ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχέσεις με την Λευκορωσία βρίσκονται ακόμα σε φάση οικοδόμησης με λιγότερο ε, προβλέψιμα αποτελέσματα. Δεδομένων των διαφορών, λοιπόν, Τώρα περνάμε σε μια επόμενη φάση μεγαλύτερη εμβάθυνση σε διάφορε ευρωπαϊκέ πολιτικέ και πρωτοβουλίε. Η ενδυνάμωση τη δημοκρατία και των δημοκρατικών θεσμών με παράλληλο σεβασμό προς ε, το διεθνές δίκαιο, η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακαιρεότητα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές για την οικοδόμηση πιο στενών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανατολικών της γειτόνων. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σημασία τη περιφερειακή σταθερότητα και τη Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσει πιο προδραστικά και να λάβει ηγετικό ρόλο στην ε, στήριξη και διευκόλυνση των ειρηνικών λύσεων ε, σε υπάρχουσε συγκρούσει. Αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκλημένοι, η ανατολική εταιρική σχέση χρειάζεται περισσότερη πολιτική στήριξη για την επόμενη δεκαετία της ύπαρξής τη που θεωρώ ότι θα φέρει ακόμα πιο απτά αποτελέσματα και αμοιβαία επιτεύγματα. Ω εισηγητή για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, χαίρομαι ιδιαίτερω που στη σημερινή ακρόαση έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εξεχουσών προσωπικότητων που έχουμε προσκαλέσει για μια ανταλλαγή απόψεων. Προσμένω λοιπόν να ακούσω πολλά και ενδιαφέροντα, να έχουμε μια ε, παραγωγική ανταλλαγή απόψεων που θα μας βοηθήσει να προετοιμάσουμε τις εκθέσει μας προ όφελο ημών και των χωρών της Ανατολική Εταιρικής Σχέσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γερασίμτσου. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για την κατάσταση στην ε, Ουκρανία, τη Λευκορωσία και την Δημοκρατία της Μολδαβίας που αποτελούν όλες μέρες του προγράμματος γειτονίας. Όμως καταρχάς ήθελα να θέσω το βασικό ερώτημα. Ποιος είναι ο βασικός σκοπός της Ανατολικής Γειτονίας και εδώ πρέπει να πω ότι η πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαράχτηκε ως ένα τρόπο για να θέσουμε κοινέ προτεραιότητε μαζί με του γείτονέ μα που να επικεντρώνεται λιγότερο στην περισσότερη διεύρυνση και στο να έχουμε σταθερότερε σχέσει περισσότερο μαζί του. Οι Βρυξέλλε έχουν πολλού πολιτικού και οικονομικού πόρου για να δημιουργήσουν ε, ένα χώρο δημοκρατία και ασφάλεια γύρω από την ε, Ένωση. Και αυτό για να υπάρξει μια ζώνη τέτοιου, γεωγραφική ζώνη τέτοιου τύπου. Έξι είναι οι χώρε, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία, όπου έχει εφαρμόσει μια πολιτική προσέγγιση για την Ανατολική Γειτονία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηριχθεί και από τη Σουηδία και την Πολωνία αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ανατολική Γειτονία με θεματικές πλατφόρμες για τις σχέσεις με τις ε, έξι αυτές χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν κοιτάξει την καλή διακυβέρνηση την ε, σωστή διακυβέρνηση ε, τον εκδημοκρατισμό και την δυνατότητα να υπάρξει ένα καλό πολιτικό πλαίσιο. Ωστόσο, η κοινωνία, ιδίω στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ε, παραπονιούνται ότι λείπει η συνιστόσα της ασφάλειας. Εδώ Υπάρχει η ήπια προσέγγιση και η πιο αυστηρή προσέγγιση στην ασφάλεια. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολύ όρεξη να εμπλακεί σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας ε, και προστασία είναι από του πυλώνε που είναι από του πιο αδύναμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη. Όμω, σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προχωρήσουμε με την Ανατολική Γειτονία, θεωρούμε ότι τα προγράμματα ασφάλεια πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Επίση, έχουν προωθηθεί πολλέ μεταρρυθμίσει στι χώρε αυτέ. Οι έξι χώρε έχουν αυξήσει το επίπεδο εκδημοκρατισμό και προόδου στην ευρωπαϊκή διαδρομή του. Επίση, υπάρχουν διαφορετικοί αντικρώμενοι ε, στόχοι στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιε φορέ. Έχουμε τις ε, συμφωνίε σύνδεση με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την ε, Λευκορωσία που υπέγραψαν τέτοιε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και χώρε όπως η Ερμενία και η Λευκορωσία, συγγνώμη, η οποία είναι πολύ πιο κοντά ακόμη στην ε, Ομοσπονδία της Ρωσίας. Η Ρωσία ακόμη λέει ότι είναι μέρος της δικής της σφαίρας επιρροής οι χώρες αυτές αλλά υπάρχουν και άλλοι στην ε, περιοχή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλοι παράγοντες. Η Κίνα είναι όλο ένα και πιο δραστήρια και συζητάμε χώρε τη περιοχή. Τώρα, αν δούμε τα πράγματα χώρα προ χώρα, η Λευκορωσία είναι μεταξύ των ε, έξι αυτών χωρών που πολιτικώ ε, είναι εγκύτερα στην ε, Ρωσία και πιο απομακρυσμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρωσική επιβολή επηρεάζει τα εσωτερικά πράγματα τη χώρα και την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων. Δεν περιμένουμε σημαντικέ πολιτικέ αλλαγέ στο προσχέ μέλλον. Η Λευκορωσία προσπαθεί να διατηρήσει την κυριαρχία της και την ανεξάρτητη εξωτερική της πολιτική, όμως ε, εξορισμού πρέπει να ε, δεχτεί τις επιλογές της και να τις ε, συσχετίσει με τις ρωσικές προτεραιότητες όπως το δικαίωμά της για να ψηφίζει για θέματα σχετικά με την Ουκρανία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Είναι και θέμα εδαφικής προστασίας. Ε, και των όσων προστάζει το διεθνέ δίκαιο. Η Λευκορωσία λοιπόν στο εξωτερικά στηρίζει τη Ρωσία. Τη συζήτηση αυτή την έχουμε επανειλημμένω με Λευκορώσου συναδέλφου σε πολλά επίπεδα και στο επίπεδο τη κοινωνία των πολιτών και κάθε φορά που θέτουμε το ερώτημα απαντούν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γι' αυτό α μιλήσουμε για οικονομία. Υπ' αυτές τις συνθήκες ε, είναι σχετικά πιθανό η Λευκορωσία να έχει τη διάθεση να αλλάξει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και να ακολουθήσει μια ευρωπαϊκή διαδρομή. Ε, Απέναντίας υπάρχει πιθανότητα η Ρωσία να ενισχύσει τη θέση της ε, στη Λευκορωσία παρά τις προσπάθειες του Μίνσκ να διαφοροποιήσει τις σχέσεις του μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Η Λευκορωσία έχει δεχτεί τη συμμετοχή της στην Οικονομική Ένωση της Ευρασίας και η Ρωσία τα ρωσικά μάλλον σχέδια είναι μια εναλλακτική λύση στην Ευρωπαϊκή Ένταξη. Η Ρωσία μπορεί ε, σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσει την οικονομική πολιτική και ε, ε, στρατιωτική μόχλευση που έχει στην Λευκορωσία για να αντιδράσει στις δυτικές βλέψεις. Είναι λοιπόν η Λευκορωσία στην αποκλειστική ζώνη συμφερόντων της Ρωσίας ή τουλάχιστον έτσι ε, την αντιμετωπίζει η Ρωσία και προσπαθεί να ε, απεμπολίσει κάθε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει επιρροή εκεί. Δηλαδή μπορεί να γίνει ό,τι δεν αντίκειται στις ρωσικές φιλοδοξίες και προσδοκίες. Από την πλευρά τη Λευκορωσία, είτε μιλάμε για κοινωνία των πολιτών, είτε πολιτικών ελίτ, είτε ε, Λευκορώσων βουλευτών, η οικονομική συνεργασία ενδιαφέρει, αλλά τίποτα περισσότερο. Η κατάσταση είναι διαφορετική με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Οι ψηφοφόροι εξέφρασαν ρητό στην βούλησή του να στηρίξουν τι προευρωπαϊκέ πολιτικέ, τι ε, φιλευρωπαϊκέ μάλλον πολιτικέ ελίτ, στι ε, πρόσφατε εκλογέ και έτσι υπογράφτηκαν συμφωνίε σύνδεση οι οποίε επέτρεψαν να γίνει σημαντική πρόοδο στον εκδημοκρατισμό, τον εξευρωπαϊσμό και τι πολιτικέ μεταρρυθμίσει. Με ένα νέο προσανατολισμό προ τα ευρωπαϊκά μοντέλα και πρότυπα. Υπάρχουν και σοβαρέ ε, παρενέργειε, διότι ακόμη και αν οι αποσχιστικέ τάσει έχουν μετατρέψει το καθεστώ ε, στην Δημοκρατία τη Μολδαβία σε μια φιλευρωπαϊκή προσέγγιση στα οικονομικά και την Συμφωνία Σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αλλά υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ε, η παγωμένη σύγκρουση στη Μολδαβία από το 1992 περιορίζει τις δυνατότητες ε, συνεργασίας ασφάλειας με τη Μόσχα. Η Ρωσία είναι και πηγή προκλήσεων. Και στη Μολδαβία υπάρχουν μετατοπίσεις είτε προς τις φιλορωσικές δυνάμεις είτε προς τις φιλευρωπαϊκές. Ο πρόεδρο αρχηγός τη βουλή και αρχηγός τη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, α πούμε, είναι υπέρ των Ρώσων. Θα δούμε όμω τι θα γίνει και με τι εκλογέ φέτο, όταν η Δημοκρατία τη Μολδαβία ε, θα περάσει σε προεδρικέ εκλογέ. Υπάρχει πιθανότητα ο νέο πρόεδρο που θα πάρει την πλειοψηφία, ο πρόεδρο μάλλον που τώρα έχουν, να ενισχύσει τη θέση του παίρνοντα την πλειοψηφία. Όπω βλέπετε λοιπόν, η Συμφωνία Σύνδεση δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα εφαρμόζεται αμετακλήτω και χωρί ε, καθυστερήσει στην Μολδαβία. Υπάρχουν και, υπάρχει και σοβαρά επίπεδο διαφθορά στι πολιτικέ ελίτ ε, και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι φιλευρωπαϊκέ ελίτ είναι εμπλεγμένε σε τέτοιε υποθέσει και αυτό ε, βεβαίω δεν επιτρέπει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών αυτών απρόσκοπτα. αμέτρητα σκάνδαλα που έχουν δυσκολέψει την πορεία ευρωπαϊκής ένταξης. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις και ο ρυθμός ε, υλοποίησης τους έχουν απογοητεύσει. Στην Μολδαβία έχουν αποτύχει οι σχετικές προσπάθειες. Οι τάσεις παραμένουν φιλορωσικές και όπως είπα, προεδρικές εκλογές θα δημιουργήσουν πολλά θα, νέα στοιχεία, θα μας δώσουν πολλά νέα στοιχεία. Επίσης η υβριδική επίθεση κατά της Μολδαβία, της Μολδαβίας, ε, ε, είναι κάτι που ε, έχει βοηθήσει τη ρωσική προπαγάνδα να βάλει στις χώρες αυτές μια ετικέτα ότι είναι αποτυχημένα κράτη και χρειάζονται την προστασία της. Κάτι άλλο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι οι τάσει τη ε, απελευθερωμένη πολυμερού προσέγγιση των οικονομικών κύκλων τη ψηφιακή επανάσταση και των ε, τεκτονικών αλλαγών που θα προκαλέσουν και είναι αισθητά σε όλε τι ε, χώρε τη Δυτική Ευρώπη, τη Κεντρική και τη χώρα τη Ανατολική Γειτονία. Μέχρι το τέλο του Φεβρουαρίου, μαζί με γερμανικά καταπιστεύματα και επίσης δυνάμεις από την Πολωνία και τον Περολίνο θα κοιτάξουμε ε, πώς θα διαμορφωθεί σχετική μελέτη και τα πορίσματά της. Ο εκδημοκρατισμός λοιπόν και ο εξευρωπαϊσμός των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας έχουν ακόμη πολλά ε, στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν και υπάρχουν ε, κριτήρια που πρέπει να συμπληρωθούν ακόμα για να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διαδρομή. Βεβαίω, ε, πριν ξέρω ότι δεν είναι κάτι άμεσο η μελλοντική διεύρυνση και οι συνομιλίε διεύρυν... Ε, ένταξη, όμω θα πρέπει να υπάρξει ε, έστω μια τέτοια προοπτική θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη και την ε, προσέγγιση της αυστηρής ασφάλειας πέραν της ήπιας για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας βάσει των όσων κάνει η Ρωσία. Η αρχική ιδέα της Ανατολικής Γειτονίας ήταν αυτή η γεωγραφική ζώνη προστασίας. Μην το ξεχνάμε αυτό μην αφήσουμε τις έξι αυτές χώρες να γίνουν ε, πηγή αστάθεια κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δώσουμε και προσοχή στην ενδυνάμωση και την σταθεροποίηση του περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στις χώρες της περιοχής. Η ευρωπαϊκή ένταξη είναι ένα θέμα επιβίωσης για τους πολίτες εκεί. Θα θέλουν πάντοτε την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών τους και θα προτιμούν να είναι σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική επικοινωνία και την ε, πρόοδο των χωρών αυτών. Η Μολδαβία παραμένει παρόλα αυτά ευάλωτη στις ρωσικές ε, ε, κινήσεις. Έγινε μια μελέτη για τις φυλακές στις περιοχές αυτές που κάλυπτε τις χώρες της Βαλτικής, του Βίσεγκραντ και τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και μεταξύ όλων αυτών η Μολδαβία είναι ο αδυναμότερος κρίκος. Επίση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά στι περιοχέ αυτέ, στην Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία. Η ρωσική επιρροή στι χώρε αυτέ ε, στοχεύει του πόρου των χωρών αυτών και κοιτάζει η Ρωσία πώ θα του παρασύρει στη διαφθορά. Ε, είναι κάτι που ισχύει ιδίω για την Ουκρανία και τη Δημοκρατία τη Μολδαβία. Το βασικά ζητήματα λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη νέα δεκαετία είναι πιστεύω, τα ζητήματα της ασφάλειας, της καταπολέμησης, της προπαγάνδας, της διαφθοράς και της υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών. Ε, σας ευχαριστούμε για την άποψή σας και τα όχι πολύ αισιόδοξα σχόλια για την κατάσταση στην περιοχή. Πάντως, ε, μας δώσετε κάποιες συστάσεις και συμπεράσματα για το πώς θα ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τώρα, ο συνάδελφος από τη Γεωργία, ο κύριος Κακάτσια. Έχετε 12 λεπτά κύριε καθηγητά για να μας παρουσιάσετε τη δική σας παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μετά τον φίλο Σεργέη Γεράσιμτσουκ εγώ θα δώσω έμφαση περισσότερο στα άλλα τρία μέλη, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και τη Γεωργία, τα άλλα τρία μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Πρώτα όλα όμως ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Όταν μιλούμε για την περιοχή, τι εννοούμε. Γιατί για μας έχουν λάβει χώρα κάποιες αλλαγές στην περιοχή. Γιατί ε, ο Νότιος Κάφκασος ε, ήταν τμήμα της περιοχής. Στη δεκαετία του 90 έτσι το θεωρούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά όμως τη θέσπιση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δεν είναι πια σαφές αν ο Νότιος Κάφκασος είναι υποπεριοχή, είναι τμήμα της ε, ευρύτερης περιοχής ή μια γκρίζα ζώνη, ένα απομονωμένο τμήμα. Τι είναι ακριβώς, ποιο είναι το καθεστώς του καυκάσου Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Τι ισχύει για τον Νότιο Κάφκασο. Και όταν μιλούμε για τον Νότιο Κάφκασο, η Γεωργία έχει συνάψει μια σύμφωνια σύνδεσης και πριν από αυτό φαινόταν ότι ήταν μια διαλυμένη περιοχή και όταν εννοούσα διαλυμένη εννοώ πολιτικά ε, γιατί ιστορικά και οικονομικά ήταν μια νέα περιοχή και αντιλαμβάνομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δικασία του 90 μιλούσε για νέα περιοχή. Τώρα όμως ε, οι τρεις χώρες, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Γεωργία έχουν λάβει διαφορετικές ε, κατευθύνσεις της πολιτικής τους. Οπότε είναι πιο δύσκολη η διαπεριφερειακή συνεργασία. Και ενώ η Γεωργία προσπαθεί να είναι πιο κοντά για προφανείς λόγους ε, στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, άλλες δύο χώρες του Νοτιού Καυκάσου έχουν διαφορετικές πορείες εξωτερικής πολιτικής. Ό,τι αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, έχουν ε, διαφορετικές ε, καταστάσεις τρεις χώρες. Μετά το 2018 και την Βελούδινη Επανάσταση στην Αρμενία έχουμε μια νέα όθηση για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και η νέα ηγεσία της Αρμενίας προσπαθεί να διεξαγάγει κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουν προβλήματα με το κράτος δικαίου και κάποιες περιπτώσεις μικροδιαφθοράς. Έχουμε θεμελιώδεις αλλαγές και στην πολιτική συμπεριφορά και στο δημόσιο λόγο, κάτι που είναι θετικό και παρά τις προκλήσεις αυτές, γενικώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωση στην περιοχή και συνεργασία με την Αρμενία και ελπίζω να συνεχίζετε να στηρίζετε τις αρμενικές μεταρρυθμίσει. Ό,τι αφορά το Αζερβαϊτζάν, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει αρκετά τοξικές τελευταία. Ε, κυρίως ε, η ευρωπαϊκή στήριξη αφορά τεχνικά, ανθρωπιστικά, οικονομικά και ενεργειακά θέματα, θέματα συνεργασίας. Ενδιαφέρει ε, το Αζερβαϊτζάν λιγότερο ε, ε εταίρος για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και φαίνεται ότι το Μπακού δίνει περισσότερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση και τι σχετικέ μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση, στην ενέργεια και τι υποδομέ μεταφορά και όχι τόσο στι δημοκρατικέ διαδικασίε. Γι' αυτό είναι και δύσκολε οι διμερεί σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά τη Γεωργία, η Γεωργία εξακολουθεί να είναι ο βασικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Υπάρχουν όμω κάποιε προκλήσει, μια και έγιναν κάποιε παλιδρομήσει πέρυσι και πρόπερσι, το 2018 και 2019, ε, προεδρικές εκλογές, αποτυχημένες εκλογικές μεταρρυθμίσεις, οι βίες καταστολές διαδηλώσεων, ε, η πόλωση και η πολιτικοποίηση της δικαστικής διοίκησης, η άτυπη διακυβέρνηση, ασύμετρη, ε, οικονομική, οικονομική και διοικητική πόρη, σημαντική επιρροή των μεγάλων ΜΜΕ στην Γεωργία και επίσης ε, ένα σημαντικό, μια σημαντική δοκιμασία, λιδία-λίθο δηλαδή για τη δημοκρατία που θα περάσει του χρόνου στις προεδρικές εκλογές του 2020 η Γεωργία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και εκλογές στο Αζερβαϊτζάν. Τώρα τι να περιμένουμε από εκεί, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά καλύτερα να επικεντρωθούμε ε, την εποχή μετά τα αποτελέσματα. Θα δούμε, βλέποντα και κάνοντα με τι εκλογέ. ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο, και οι τρει χώρε, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Γεωργία, προσπάθησαν να σφαιριλατήσουν σχέσει σε διαφορετικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μάλιστα, η ΣΕΠΑ με την Αρμενία, η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση ενισχύθηκε το 2018, αλλά δεν περιλαμβάνει και σφαιρική και σε βάθο ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Μάλιστα η Ερμηνεία είναι μέλος και της Ευρωσιακή Ένωσης υπό τη ρωσική πίεση, κάτι που παρεμποδίζει την βαθύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό δεν επηρεάζει το εμπόριο τη Αρμενία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο μείζον εμπορικό εταίρο Τη Αρμενίας και πάροχος χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης. Ό,τι αφορά το Αζερβαϊτζάν, οι συμβατικέ σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να στηρίζονται στη Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία του 1999. Είναι σημαντικότερο ενεργειακό και εμπορικό εταίρο ε, του Αζερβαϊτζάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αζερβαϊτζάν παρέχει 5% του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Οι επικείμενε εκλογέ θα έχουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, Έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία σφαιρική και σε βάθο ε, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών από το 2014. Η εφαρμογή τη όμω είναι δύσκολη, επίπονη και επώδυνη διαδικασία και πολύ δαπανηρή για την γεωργία. Είχαμε κάποιε θετικέ εξελίξει εκεί, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιε προκλήσει σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι δυστυχώς παρόλο που έγινε μια απόπειρα και από τις δύο πλευρές με βάση τις στατιστικές του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας. Ε, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εταίρος που ε, έχει το 53% του ε, εμπορίου με τη Γεωργία, ενώ το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 22% μόνο. Οπότε θα πρέπει να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωργίας. Υπάρχει χώρος εκεί. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, την σταθερότητα και την ασφάλεια, εδώ έχουμε μια ε, παγωμένη σύγκρουση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Μακροχρόνια σύγκρουση και μάλιστα κάτι τέτοιο υπονομεύει την ε, σταθερότητα της περιοχής και ε, εδώ είναι περιορισμένος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα βέβαια είπα έχει παραπευθεί στον ΟΑΣΕ το Αζερβαϊτζάν θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ παθητικό παράγοντα που δεν τον υποστηρίζει στην περιοχή, ενώ η Ρωσία χειραγωγεί και την αρμενική και την αζερβαϊτζανική κοινωνία, την αζέρικη κοινωνία, πουλώντα όπλα και στι δύο πλευρέ, κάτι που δυσχεραίνει την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την Γεωργία, η ασφάλεια και σταθερότητα της Γεωργίας υπονομεύεται από την διαδικασία της συνοριοποίησης, όπως τη λέμε, από τη Ρωσία. Έχουμε και την κατοχή της Απχαζίας και της Νότιο Οσετίας και σίγουρα θα είναι η κυριότερη πρόκληση στο μέλλον η ασφάλεια για τη Γεωργία. Και παρόλο που έχει ένα δίλημα ως προς τη Ρωσία για την ασφάλεια η Γεωργία, εξακολουθεί να κρατά του ισχυρού στρατιωτικού δεσμού που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μάλιστα την αποστολή επιτήρηση Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008, σημαντικός σταθεροποιητικό παράγοντας. Και επίση η Γεωργία συμμετέχει σε επιχειρήσει ασφάλεια και άμυνα Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει στείλει στρατεύματα στο Μάλι και σε άλλε αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημαντικότερη πρόκληση που έχουμε εδώ αφορά τη δημοκρατία στη Γεωργία. Και πλησιάζοντας τα συμπεράσματα θα πρέπει να ενισχύσουμε την, την πίεση εκδημοκρατισμού στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε σημαντική επιρροή, κυρίως στη Γεωργία και εν μέρει και στην Αρμενία. Το 2020 θα είναι σημαντικό για τη δημοκρατική εξέλιξη και τη μεταρρύθμιση της Γεωργίας. Υπάρχει κίνδυνος βέβαια παλινδρόμησης λόγω της εσωτερικής αστάθειας στη Γεωργία. Και μάλιστα ε, αν αποκοπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφήσει ελεύθερο χώρο και περιθώριο στη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα για να προβούν σε χειραγώγηση και ελιγμού στην περιοχή. Επίση, θα πρέπει να αναβαθμιστούν ε, οικονομικέ και στρατηγικέ συμμετοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέδια υποδομών που θα συνδέουν την Κασπία με την Ευρώπη και καλό θα ήταν ε, να διευκολυνθεί η Γεωργία να εφαρμόσει κάποια πιο δαπανηρά τμήματα τη ε, ε, ει βάθο και σφαιρική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, κυρίως για την εφαρμογή των προτύπων. Ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή σε αποστολέ, ε, είναι ανεπαρκή ακόμη. Θα πρέπει να αναβαθμιστούν και ίσω να ξεκινήσει ένα είδο συμφώνου σταθερότητα τη Ανατολική Εταιρική Σχέση που θα συμπεριλαμβάνει και το Νότιο Κάφκασο. Αλλά αυτό είναι αντικείμενο ίσω ξεχωριστή συζήτηση. Θα ήταν μία από τι ιδέε όμω που θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ποια είναι τα μαθήματα τώρα. Σίγουρα μια περιφερειακή προσέγγιση χρειάζεται, αλλά μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση για τα προβλήματα. Χρειάζεται πιο ηγετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόσθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίση να προωθηθεί η ταυτότητα τη Ανατολική Εταιρική Σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για να γίνει κάτι τέτοιο θέλουμε ένα νέο δικό χάρτη. Σε ό,τι αφορά τι περιφερειακέ πρωτοβουλίε για το Νότιο Κάφκασο, Ίσως θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο διμερείς σχέσεις και κάποιες κοινέ ομάδες ε, παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει τους θεσμούς, τη διακυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και όχι μόνο την κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας για να ενισχύσετε τις μεταρρυθμίσεις εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου, κυρίως στη Γεωργία, προσφέροντα πιο εξατομικευμένε διμερεί λύσει και στηρίζοντα ε, την κοινωνία των πολιτών. Η σταθερότητα είναι πολύ χρήσιμη, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια εταιρική σχέση που θα δράζεται στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Εν κατακλείδη, σημαντικό είναι να επενδύσουμε στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε καθηγητά για την περιγραφή της κατάστασης αυτές τις τρεις χώρες και για τις προτάσεις που μας δώσατε για τη βελτίωση της κατάστασης. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σάρη. Έχετε 12 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προηγούμενους ομιλητές που περιέγραψαν ε, την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ορισμένες από τις ε, βασικές προκλήσεις ε, στην περιοχή σήμερα. Εγώ σήμερα θα ήθελα να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Τι πρέπει να γίνει, πώς το πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα πρέπει να προσαρμοστεί, ούτως ώστε να είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει φυστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Η παρουσίασή μου βασίζεται στην ανάλυση που κάναμε με τον συνάδελφο ε, Στάνισλαβ Σεκριερού πέρυσι και θα ήθελα να προτείνω τρεις ε, βασικές άγουσες για την ε, επικαιροποίηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης για την επόμενη δεκαετία. Μπορείτε να βρείτε και αντίτυπα της ανάλυσης μας εδώ στα δεξιά. Το πρώτο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε ε, την νοοτροπία και τρόπο σκέψη μα σε ό,τι αφορά την Ανατολική γειτονία. Γιατί η περιοχή αυτή έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, α πούμε. Είναι πολύ δυναμική και πολυκεντρική περιοχή ή πολυπαραγωγική. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τι χώρε τη Ανατολική Εταιρική Σχέση ω ε, ε, κράτη στόχου ή σαν ένα project φιλανθρωπίας. Τα τελευταία χρόνια πολλές από αυτές τις χώρες έχουν λάβει ένα καθεστώ πραγματικού εταίρου και συμβάλλουν σημαντικά στο κοινό θεματολόγιο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εποφελείται από την Ανατολική Εταιρική Σχέση και οι οικονομίες των χωρών μας. Ε, παρέχει επιχειρηματικές δυνατότητες, αυξάνει ε, την πολιτική θέση και το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύεται και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όλα αυτά θα πρέπει να τα επικοινωνούμε με καλύτερο τρόπο και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολύ συχνά κάπως ε, μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχουν και τρίτες χώρες όπως ε, η Κίνα, η Τουρκία και οι χώρες ε, του Περσικού κόλπου που έχουν αυξήσει τις διπλωματικές και οικονομικές τους προσπάθειες και την επιρροή τους σε αυτές τις χώρες. Δεν πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε μόνο τη Ρωσία και τον ρόλο και την επιρροή που έχει, αλλά και άλλες δυνάμεις. Κάποιες φορές οι αξίες ε, και μέθοδοι τρίτων χωρών δεν αντιστοιχούν στις δικές μας. Όμως, εν γέννη, οι αυξανόμενες εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες αυξάνουν την οικονομική ανθεκτικότητα των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και αυτός είναι στόχος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες να οικοδομήσουμε ισχυρότερες εταιρικέ σχέσεις ε, με δυνάμεις που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς, καθώς και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα και φορείς. Έχουμε για παράδειγμα τη συνάντηση ε, των πρεσβευτών των χωρών G7 στην Ουκρανία. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να διοργανωθεί και σε άλλες ε, χώρες τη Ανατολική εταιρική σχέση. Τρίτον, υπάρχουν αυξανόμενε διασυνδέσεις μεταξύ ε, των χώρων της Ανατολικής και της Νοτίου εταιρικής σχέσης. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα εξετάζουμε αποκομμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα χρειάζεται μία ε, σφαιρική οπτική της ε, κατάστασης και μία ολοκληρωμένη και σφαιρική στρατηγική για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, και στην Ανατολή και στον Νότο. Μπορούμε στη συνέχεια να αναφέρουμε λεπτομέρειες ως προς αυτό. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο πυλώνα επικαιροποίηση των πολιτικών μας. Πρέπει να βελτιώσουμε τις πολιτικές για την υποστήριξη των ναι, μεταρρυθμίσεων στην Ανατολική Κεντρική Σχέση. Χρειαζόμαστε έναν ε, συνδυασμό κινήτρων και ε, κριτηρίων αρεσιμότητας. Αλλά πάνω απ' όλα να βελτιστοποιήσουμε ε, τις στρατηγικές μου για να αντιμετωπίσουμε μας για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια που προκύπτουν με έναν ε, ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο για να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον. Για παράδειγμα, κάποιες φορές οι πολιτικές ελίτ καθυστερούν και κολυσιεργούν. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει να εφαρμόζουμε τη λεγόμενη ευφυή αιρεσιμότητα. Για παράδειγμα, να ε, επαναδιοχετεύουμε ορισμένα κονδύλια σε φορεί τη κοινωνία των πολιτών ή άλλους φορείς της χώρας. Στη Μολδαβία ήδη έχουμε δει ε, πολύ επιτυχημένα πειράματα σε αυτή την προσέγγιση. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες ε, κοινωνικές ομάδες ε, που διστάζουν και είναι καχύποπτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πραγματικά να αποταθούμε στις ε, πλέον επιφυλεκτικές ομάδες και να προσπαθήσουμε να τις πείσουμε. Εν γέννη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευρύνει το φάσμα των εταίρων τη στις ε, χώρες της Ανατολικής σχέση. Η κοινωνία των πολιτών πάντα υπήρξε ισχυρό σύμμαχό μας και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Πέραν τούτου όμως, θα πρέπει να οικοδομήσουμε πιο προδραστικά ε, δεσμούς με άλλες ε, ομάδες που θέλουν να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως είναι η νεολαία, η ομογένεια, η επιχειρηματική κύκλη και ούτω καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε επίσης να εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος ε, τον κοινωνικό αντίκτυπο των ε, σχέσεών μας. Εάν με τι μεταρρυθμίσει ε, δημιουργούνται μόνο νικητές και χαμένοι, ακόμα και η οικονομική ανάπτυξη δεν θα φέρει σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή. Πρέπει να σκεφτούμε νέα κίνητρα που θα ωφελήσουν τον απλό κόσμο την ε, πλειονότητα λοιπόν του κόσμου που δεν ανήκουν στα, ε, στις ε, αστικές μειονότητες υψηλού μορφωτικού επίπεδου που υπάρχει σε αυτές τις χώρες. Επιπλέον, η έλλειψη προόδου μπορεί να συνδέεται και με την έλλειψη γνώσεων, τεχνογνωσίας και συνδέσεων και υποδομών. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας, ισχυρότερους δεσμούς με τους επιχειρηματικούς κύκλους και θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, διασυνδεσιμότητα και ε, σε έργα υποδομών για, το, για την περιοχή αυτή. Οι επικοινωνικές στρατηγικές θα πρέπει ε, να έρθουν στην ψηφιακή εποχή. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στις αντιπροσωπείες μας στην Ανατολή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε απλά και προσιτά μηνύματα για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις χώρες και πώς Όλα αυτά ωφελούν ε, τους πολίτες. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις τοπικές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από αυτές τις ενισχυμένες ε, εμπορικές σχέσεις. Για παράδειγμα στη Γεωργία πώς ε, μπορούν εκείνοι να ε, φτάσουν, να βρουν τον δρόμο προς την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξήσουν το μερίδιό τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και να πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Και θα πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση στενότερων δεσμών προκειμένου ενδεχομένω να ενταχθούν αυτές οι χώρες ε, και στις ε, ευρωπαϊκές αγορές. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, είναι θετικό που αυξάνονται οι πορικές σχέσεις, όμως ε, οι υποδομές δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιο επίπεδο συναλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθούν οι υποδομές των χώρων αυτών και να συνδεθούν με τις ευρωπαϊκές. Είναι κύριο μέλημα για την επόμενη δεκαετία αυτό. Και ο τρίτος ε, πυλώνας ε, για το μέλλον είναι ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, τις διασυνδέσεις και αλληλοεξαρτήσεις ασφαλείας ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Υπάρχει η αντίληψη ότι όλο αυτό ωφελεί μόνο τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Πριν από μια δεκαετία θεωρούσαμε ότι τα, ε, τα μέσα επιβολής της Ρωσίας ε, στόχευαν μόνο τις χώρες αυτές. Όμως, τελικά, είδαμε ότι όσα γίνονταν τότε στην Ανατολή, μετά έγιναν και στη Δύση εκστρατείε παραπληροφόρηση, κυβερνοεπιθέσει και το καθεξής. Οι ε, προκλήσεις στον κυβερνοχώρο είναι ένα θέμα που πραγματικά θα πρέπει να εργαστούμε ε, από κοινού. Απαιτείται επίσης ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και στις ε, πρωτοβουλίες καταπολέμησης της νομοποίησης εσόδων από παράνομες πηγές. Και όλα αυτά πρέπει να αφορούν ε, πολυεπίπεδη συνεργασία σε βάθος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινέ ε, δοκιμές για τον κυβερνοχώρο και συζητήσεις με τα τρία συνδεδεμένα κράτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι τέτοιο για τη Βραζιλία, αλλά όχι για κάποια χώρα της Ανατολικής Τερικής Σχέσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντική έλλειψη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δράσουμε προληπτικά και όχι εκ των υστέρων, όπου συχνά ο οικονομικός ε, αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς και ο κίνδυνος για την ασφάλεια. Τρίτος παράγοντας, η διαφθορά θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο σε ένα θέμα που συνδέεται με την οικονομία και τη διακυβέρνηση, αλλά και με την ασφάλεια. Η διαφθορά διευκολύνει και δίνει κίνητρα για τις ε, ε, απειλές, ε, τις υβριδικές απειλές. Η καταπολέμηση διαφθοράς ανήκει σε όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Θα πρέπει λοιπόν να, δρούμε και τον, εκ των υστέρων αλλά και προληπτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Σάρη για την συνεισφορά σας για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της Ανατολικής Γειτονίας για τα ερχόμενα 10 χρόνια και παραπέρα. Ίσως κάποια στιγμή να υπάρξει και ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να ακούσουμε τώρα τον προσκεκλημένο μας από το Βίλνιους, τον κύριο Μανιώκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι του μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πάνω από 10 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, η Ανατολική Γειτονία έχει αποδείξει ότι είναι ένα βασικό εργαλείο για την συμμετοχή και την διαμόρφωση σχέσεων των Ανατολικών γειτόνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γείτονε αυτοί έχουν έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τι διευρύνσει του 2004 και 2007 και με το επίπεδο τήρηση, μάλλον με το, επί, με το επίπεδο προσδοκιών και αλληλεξάρτησης που έχουμε επιτύχει, η Ανατολική Γειτονία έχει ήδη δώσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Όμως μετά από 10 χρόνια βλέπουμε και ποιες, ποια είναι τα όρια και ποια τα αμφιλεγόμενα σημεία της πολιτικής αυτής. Και πολλές από τις ε, δυσκολίες και τις ελλείψεις είναι και τις ίδιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελλείψεις. Πρώτα απ' όλα η πολιτική στόχη της Ανατολικής Γειτονίας, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, ο εξευρωπαϊσμός, ω προ του κανόνε και τα πρότυπα, η εθνική κυριαρχία, η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη τη γειτονία. Πώ σχετίζονται όλα αυτά με του πολιτικού στόχου και τι ανάγκε των ε, γειτόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερη σύγκληση μεταξύ των συμφερόντων Ευρωπαϊκή Ένωση και των εταίρων, τους, ε, των εταίρων της είναι ε, σαφώ ένα δρόμο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Όμως κάποιες φορές ε, μπορεί αυτά τα συμφέροντα και ανάγκες να είναι αντικρώμενα μεταξύ του. Μπορεί οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να με διαθέτουν αυτά που απαιτεί η Ανατολική Γειτονία. Αυτό που κυρίως χρειάζονται και δεν μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γείτονε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ασφάλεια. Υπάρχει σοβαρό περιορισμό λόγω των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη και αποστολέ κράτου δικαίου ε, και τήρηση του κράτου δικαίου, όσο και αν είναι καλέ, δεν αρκούν. Είναι πολλά τα επίπεδα προσαρμογή που χρειάζονται ακόμα και είναι θεμητά και ευπρόσδεκτα. Υπάρχει μια πολιτική πλατφόρμα ενιαία για την ε, διαμόρφωση των χωρών αυτών που πρέπει να έρθουν πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά ακόμη και με το πρότυπο της διεύρυνσης δεν είναι αρκετά όλα αυτά για να υπάρξουν τόσα κίνητρα ώστε να πετύχουν ευρωπαϊκή ένταξη. Και μιλάμε για χώρες που έχουν περάσει σε ένα καθεστώς ε, πολιτικό που ε, ξέφυγε από τη Σοβιετική Ένωση και δημιουργεί ένα άλλο πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των γειτόνων αυτών, πρέπει να δούμε τις διαφορετικές τους φιλοδοξίες με τον σωστό τρόπο. Και να λάβουμε υπόψη και τους περιορισμούς αλλά και το τι πόρους διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξουν να υπάρξει καλύτερη στοχοποίηση του πώς θα εξισορροπηθούν οι πόροι αυτοί. Και η διαφοροποίηση πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χωρών στην Ανατολική Γειτονία. Υπάρχουν χώρες ε, μετάβασης και χώρες σύνδεσης. Ας πούμε, Είναι αντιπαραγωγικό το να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ένταξη. Θα πρέπει κυρίω να επικεντρωθούμε στα σωστά μέσα και τους πόρους. Ω προ τη διαφοροποίηση, αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον δύο κατηγορίε, δύο λογιών χώρε, ίσω και περισσότερε. Και περισσότερα σύνολα στόχων και μέσων που πρέπει να αξιοποιηθούν στην κάθε περίπτωση. Πρώτα απ' όλα έχουμε τι συνδεδεμένε χώρε τη Ανατολική Γειτονία που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση με μία από τι πολυπλοκότερε και φολιδοξότερε συμφωνίε που έχουμε ουδέποτε συνάψει με τρίτα μέρη. Στην ομάδα αυτή ανήκουν η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία αυτή τριάδα συνδεδεμένων χωρών. Μια άλλη ομάδα είναι οι χώρε χωρί συμφωνία σύνδεση, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν και η Λευκορωσία. Η Αρμενία έχει συνάψει συμφωνία που μοιάζει με αυτήν της σύνδεση. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ως ε, μια χώρα borderline μεταξύ των δύο ομάδων. Ε, στην πρώτη ομάδα όμως ξεχωρίζει η Ουκρανία ε, λόγω μεγέθους, σημασίας και το πόσο έχει εμπλακεί στην ευρωπαϊκή της πορεία είναι η μόνη μεταξύ των έξι χωρών που έχει ξεκινήσει ένα κοινό σχέδιο οικοδόμηση των κρατικών πόρων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπερνά του στόχου τη απλή εθνική κυριαρχία, σταθεροποίηση και εξευρωπαϊσμού. Ε, αυτά τα σύνολα χωρών, οι χώρε, ε, μπορούν να λειτουργήσουν ε, ομαδικά ή ξεχωριστά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ας ξεκινήσουμε από τι δύο χώρε που έχουν δημιουργήσει τι περισσότερε αμφιβολίε ω προ την αρχική συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσφορέ που του κάναμε, Λευκορωσία και Αζερβαϊτζάν. Οι χώρε αυτέ έχουν περισσότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιου τομεί όπω η ενέργεια, στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν, και υπήρξαν ε, και κάποιε θετικέ εξελίξει με την πρωτοβουλία για τα αποτελέσματα του 2020. Η ε, βασικοί στόχοι ήταν η εθνική κυριαρχία και η σταθεροποίηση. Θέλαμε να εξισορροπήσουμε λίγο την, και να αντισταθμίσουμε την επιρροή της Ρωσίας και άλλων διεθνών παραγόντων, από της Κίνας και άλλων. Θέλαμε επίσης να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες, ιδίως της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το εξής δίλημα θα πρέπει να κοιτάξει εάν θα προωθήσει κι άλλο την εθνική κυριαρχία και τη σταθεροποίηση ή τις ευρωπαϊκές αξίες, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, χάνοντας όμως εντελώς την επιρροή της, ενδεχομένως εάν αυτό δεν πάει καλά. Ως προς τη σύνδεση, οι συμφωνίες σύνδεσης είναι από τις πλέον περίπλοκες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ φιλόδοξες ως προς την ε, νομική, την νομοθετική εναρμόνιση. Οι τρεις συνδεόμενες χώρες έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κανόνων. Αλλά υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα εδώ σε σχέση με τη σύνδεση. Ένα από αυτά είναι το πώς έχει ήδη σχεδιαστεί η συμφωνία στη δημιουργία της και ένα άλλο είναι οι δυνατότητες που έχουν οι χώρες αυτές το πεδίο και το βάθος των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται από τις συνδεδεμένες χώρες ε, δεν ε, συνδυάζεται και αντιφάσκει με το τωρινό επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει οι συμφωνίες σύνδεσης να αποτελέσουν ένα πρότυπο, ένα αποτύπωμα που θα βοηθήσει τον εξεχρονισμό της Γεωργίας Μολδαβίας και Ουκρανίας και θα αποδείξει ότι το κεκτημένο μπορεί να εξυπηρετήσει και δικές τους ανάγκες, αλλά αυτό μπορεί και να αμφισβητηθεί ε, ως ε, στόχος. Επιτά, θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα των χωρών αυτών να εφαρμόσουν τους σωστούς κανόνες και αν αυτή θα είναι αποφελής για την ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να δούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει όλους τους πόρους για να συνεργαστεί και να βοηθήσει. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα απορίσματα του προ πρόσφατου προγράμματος EU Strat ε, στα πλαίσια του Horizon και το έκτο πακέτο της σύνδεσης ε, και γι' αυτό θα σας προσφέρω τη δική μου εμπειρία από τη διαδικασία σύνδεσης και την Ανατολική Γειτονία. Ε, είναι πολύ διαφορετικά αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα στις χώρες αυτές σε σχέση με το πώς παίρνουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πώς το εφαρμόζουν. Τα περισσότερα από τα κεκτημένα δεν είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και είναι και σωστό αυτό, διότι έχουν πιο επίγουσες ανάγκες για την οικοδόμηση βασικών κρατών κρατικών θεσμών, όπω στην Ουκρανία, όπου λείπει και η οικονομική ανάπτυξη και η συνιστόσα τη ασφάλεια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποφάσισε αυτό να το αντιμετωπίσει μόνο στην Ουκρανία. Η ε, μελέτη μου έδειξε ότι η μεταφορά και η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε πολλούς τομείς είναι αποσπασματική, αλλά τα έχει πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό κυρίως γιατί διαρκώς υπάρχει μια άτυπη ε, προσαρμογή στις νέες συνθήκες των συμφωνιών σύνδεσης. Δηλαδή να μειωθεί το πεδίο των ε, δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται και ε, φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποδέχεται αυτό. Είναι θετικό βέβαια αυτό γιατί βοηθά να ελαφρύνουμε το άχθος της εναρμόνισης αλλά γίνεται βάσει της διακριτικής ευχέρεια του καθενός και δεν δημιουργεί ένα ε, ομοιογενές μοντέλο. Άρα δημιουργεί και αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το πώς θα λειτουργήσουν οι σχέσεις στο μέλλον μεταξύ διαφορετικών φορέων, όπως κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων και επενδυτών. Η μελέτη ε, επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο δίνει δυνατότητες σε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που προηγουμένως ήταν πιο αδύναμε, αλλά παραμένουν κενά στο επίπεδο της υλοποίησης λόγω των χαμηλών διοικητικών επιδόσεων και των ε, ε, συμφερόντων που αναζητούν το βραχυπρόθεσμο κέρδος, όπως στην περίπτωση των ρυθμιστών ενέργειας. Η ευρωπαϊκή αιρεσιμότητα λειτουργεί για κάποιες μόνο μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τις υπαρξιακές ανάγκες των χωρών απευθείας, όπως τη μεταρρύθμιση του τομέα φυσικού αερίου στην Ουκρανία η υλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων θα γίνεται το και περιπλοκότερη. Και αυτό δείχνει ότι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων και η εφαρμογή της αιρεσιμότητας μπορεί να παραμείνουν μόνο στα λόγια. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε απευθείας αυτόν τον κίνδυνο ως προς τις συστάσεις μας. Πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα όσο και αν είναι περιορισμένα. Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ περισσότερο στη σύνδεση, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερε σχέσει αλληλεξάρτηση και συνεργασία με τι μη συνδεδεμένε χώρε. Θα πρέπει να δούμε τι γεωπολιτικού κοινού στόχου μπορεί να έχουμε. Θα πρέπει να ε, προωθήσουμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων για τις χώρες αυτές μαζί με τεχνική αερογή και κυρίως με επενδύσεις, ξένες επενδύσεις. Η μεταφορά των ευρωπαϊκών κανόνων και η υλοποίησή τους είναι κάτι που κοστίζει χρειάζεται μια πιο αυστηρή οικονομική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί αυτή την οικονομολογική προσέγγιση να την προσφέρει με έναν κοινό οικονομικό χώρο και εφόσον ανοίξει τον ε, κλάδο των υπηρεσιών λόγου χάρη. Σε συνεργασία με τις χώρες αυτές που θα είναι συνδεδεμένες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή νομίζω είναι η βασικότερη στόχη και έτσι θα μπορούσε η συμφωνία σύνδεσης και γενικότερη διαδικασία της σύνδεσης να λειτουργήσει και μάλιστα από την οικονομική σκοπιά. Εν τέλει, για να ε, δημιουργηθεί πραγματικά η σύνδεση θα πρέπει να δούμε πιο λεπτομεριακά και ε, επισταμένως τα διάφορα κεφάλαια των συμφωνιών Σύνδεση. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και τις απόψεις σας. Και όπως υποσχέθηκα από την αρχή της συζήτησης, ε, εκτός από τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες, καλέσαμε και την κυρία Άιχορστ και την κυρία Ματερνοβά Θα δώσω το λόγο πρώτα στην εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ για 10 λεπτά, την κυρία Αγγελίνα Χόρστ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξότιμη Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ε, με εντυπωσίασαν οι παρουσιάσεις σας. Δυστυχώς δεν ήμουν από την αρχή εδώ. Πάντως ήταν πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας και οι συστάσεις που κάνατε για την ε, ανατολική εταιρική σχέση και θα τις λάβουμε υπόψη και εγώ και η Κατερίνα Ματέρνοβα. Χαιρόμαστε για την παρουσία μας εδώ. Βλέπουμε ότι γίνονται πολλές ζυμώσεις και πολλές συζητήσεις και είναι σημαντικό να συγκεντρώνουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις. Και μου άρεσε αυτό που είπε η κυρία Σάρη, ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψη και νοοτροπία ε, γιατί ο κόσμος ε, μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. Δεν θα πρέπει να μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Και αυτό ισχύει και για την ανατολική εταιρική σχέση. Έχω σύντομα τέσσερα σχόλια, μια και ο χρόνος ε, είναι λίγος. Εκτιμώ ιδιαίτερως αυτή τη δημόσια ακρόαση που οργανώσατε. Έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια αναφέρθηκε η δέκατη επέτειο στι ανατολικε εταιρικε σχεσει Πολλά συνέβησαν αυτή τη δεκαετία. Σίγουρα σημειώσαμε πρόοδο με όλου του εταίρου, αλλά και γενικά στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Και διαπιστώνουμε πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Και είναι πολύ δυναμική η σχέση μα με τι χώρε αυτέ. κάτι που είναι σχετικά καινούριο και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί και σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο δέσμευση. και αυτή είναι η άποψη και της ΑΕΘ e και του υποτεκπρόσωπου. Επανειλημμένος ε, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριος Γιωζέ Μπορέλ ότι θα δώσει προτεραιότητα στην ε, ε, ανατολική εταιρική σχέση και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία και με τι έξι χώρε σε διαφορετικά επίπεδα βέβαια. Οπότε ε, ο δυναμισμό είναι σημαντικό και θα πρέπει να χαρακτηρίζει τι ε, νέε μα σχέσει. Επίση έχουμε συνάψει τι συμφωνίε και ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Πάντως οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβάλλουμε για να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση αλλά και πολιτική σύνδεση. Και σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα της κυρία Σάρη, σίγουρα θα λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρατε κατά την προετοιμασία της επόμενης διάσκεψης κορυφής και υπάρχει και το σημαντικό πολιτικό στοιχείο. Χρειάζεται πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα και οι επικεφαλής των γραφείων μας σε όλες τις πρωτεύουσε ε, έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο δράσης από ό,τι πριν από μία δεκαετία και συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα και στο πολιτικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φυσικά αυτό γίνεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και εδώ έχει νόημα και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και είχαμε πρόσφατα κάποιες πολιτικές κρίσεις και κάποια ζητήματα με τις επιμέρους χώρες και εκεί διαπιστώνουμε ότι όταν συνεργαζόμαστε πολιτικά μπορούμε να βοηθήσουμε είτε στην αποκλιμάκωση είτε στην διατύπωση επικοδομητικών προτάσεων για βελτίωση. Πάντω όλοι οι μηχανισμοί που έχουμε επί τόπου και όλα τα εργαλεία που έχουμε και τα γνωρίζει από την καλή και από την ανάποδη όλα διεξοδικά η Κατερίνα, τα αξιοποιούμε όλα αυτά τα μέσα που έχουμε. Σίγουρα πάντως θα πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας εκεί και έχουμε ευτυχώς ένα πλαίσιο. Αν δεν το είχαμε θα έπρεπε να το κατασκευάσουμε τώρα. Πάντως έχουμε ένα πραγματικά στενερό, σταθερό πλαίσιο συνεργασίας και με τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Και βλέπουμε ότι αποφέρει καρπούς και για τους ε, πολίτες. Αυτό το επισήμανε και ο ύπατος εκπρόσωπος και το κάνει συστηματικά σε κάθε ευκαιρία. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε λοιπόν, τα ωφέλη αυτό το πλαίσιο. Και βλέπουμε και κάποια θετικά αποτελέσματα και είχαμε και ένα πολύ καρποφόρο γύρο διαβουλεύσεων το τελευταίο εξάμεινο, διαρθρωμένο διάλογο με τεράστια συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα Κοινωνία των πολιτών, κυβέρνηση από διάφορους φορείς και παράγοντες, από εμπειρογνώμονες και θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την επόμενη διάσκεψη κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο. Αυτή η Προσέγγιση όμως από τη βάση προς την κορυφή και το να οικειοποιηθούν τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενες χώρες είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά ε, το αν θα είναι επιτυχής η πολιτική αυτό θα κριθεί από τους πολίτες που είναι οι άμεση δικαιούχοι αυτής της πολιτικής και παραλήπτες. Αυτοί θα πρέπει να μας κρίνουν. Πάντως έχουμε σημειώσει πρόοδο. Έχουμε τώρα το θεματολόγιο για την εποχή μετά το 2020. Πάντως όλα τα στοιχεία που αναφέρατε, σχεδόν όλα. Ε, κάποιες χώρε βέβαια έχουν διαφορετικές ίσω αλλά σε τελική ανάλυση θέλουμε και τις 27 χώρε στο πλευρό μας. Και ζητούμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε και οι θέσει στο Συμβούλιο να μας βοηθήσουν και να προαγάγουν αυτή τη συνεργασία μεταξύ μας. Και σίγουρα στο Συμβούλιο εν ώψη και της διάσκεψης κορυφής ε, θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Μιλήσατε για συμπερίληψη, για σύνδεση, για αποφυγή αποκλεισμών, για διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολιτικά θα δώσει το στίγμα της και η διάσκεψη κορυφής. Φυσικά θέλουμε και εμβάθυνση και να δούμε ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει διαφορά και μιλήσαμε για την ψηφιοποίηση, τις κλιματικές αλλαγές. Όλες αυτές ε, είναι νέες και νέες προτεραιότητες και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τις έξι χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και για αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ματέρνοβα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Αντζελίνα για τα καλά της λόγια αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, χαίρομαι ιδιαίτερος για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ε, εμπειρογνώμονες καλεσμένους σας. Κατάγραψα ιδιαίτερα τα σχόλια του κύριου Μανιώκας, γιατί πραγματικά έχουμε πολλές κοινέ απόψεις και σκέψεις. Και θα έρθω σε αυτά σε λίγο. Από πού ξεκινάμε. Η Ευρωπαϊκή ε, Ανατολική Εταιρική Σχέση ξεκίνησε μετά την ε, επίθεση στη Γεωργία το 2009 σε ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο. Και τώρα, ε, κατά τον εορτασμό της 10ης επαιτίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ατενίζουμε το μέλλον, την επόμενη δεκαετία που θα λάβει χώρα σε ένα ακόμη πιο περίπλοκο ίσως πολιτικό πλαίσιο. Πάντως, η ο γεωπολιτικός ανασχηματισμός και η ανακατα... ανακατάταξη της σχέτησης δυνάμεων στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά και υπάρχει ισχυρή δέσμευση του Συμβουλίου αλλά και των ε, χωρών εταίρων για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής της ανατολικής εταιρικής σχέσης γιατί είναι πολλά τα ωφέλη της, όπως είπε και η Αντζέλινα Αιχόρστ. Για να δούμε όμως από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, τι έχουμε καταφέρει. Και δεν θα μιλήσω για το α ή β σχέδιο και πρόγραμμα. Θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα σημεία που δείχνουν την πρόοδό μας. Πρώτον, έχουμε τρία συνδεδεμένα μέλη με τις προκλήσεις που αυτό περιλαμβάνει. Ε, τρεις χώρες όμως που έχουν συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπλοκες και σύνθετες συμφωνίες, περίπλοκες με όλη τη σημασία της λέξης, μερικοί εμπειρογνώμονες είπατε ότι ήταν περισσότερο βάση των καλύτερων πρακτικών και όχι, δεν ανταποκρινόταν ε, με τις συγκεκριμένες χώρες. Και όντως δεν έχουμε εξατομικευμένες συμφωνίες απόλυτα, δεν προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι συμφωνίες συντάχθηκαν σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο και με την προσδοκία ότι ήταν ο προθάλαμος της ένταξης και υπήρχε προσδοκία ότι η υιοθέτηση αυτών των συμφωνιών και των αντίστοιχων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων θα έκανε ένα βήμα προ τη διεύρυνση. Ήταν πολύ διαφορετική λοιπόν η πολιτική προτεραιότητα, ε, πραγματικότητα που χαρακτήριζε τη σύνταξη των συμφωνιών. Και μερικέ φορέ δεν κοιτάμε τι υποσημειώσεις και τα μικρά γράμματα, γιατί η πολιτική σημασία τη σύναψη συμφωνία σύνδεση με το συστατικό και τη σφαιρική και σε βάθο ε, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ήταν ένα πλαίσιο με πολλές λεπτομέρειες. Πάντως, στη δεκαετία βρήκαμε τρόπους να αντισταθμίσουμε αυτή την υπερβολική περιπλοκότητα και θα ήθελα να σας δώσω τρία συγκεκριμένα ή τέσσερα παραδείγματα για το πώς τα καταφέραμε. Γιατί στην περίπτωση της Ουκρανίας το καταφέραμε και θεσμικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν αφιερώσαμε μεγάλες προσπάθειες, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, για να επαναπροσανατολίσουμε την ενίσχυση, όχι από τα όχι από, στα προγράμματα, αλλά για να στηρίξουμε ε, σφαιρικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Κάτι που γίνεται πιο συστηματικά στις συνδεδεμένες χώρες. Γιατί όσο λιγότερη δέσμευση έχουμε και λιγότερη βοήθεια, τόσο λιγότερα προγράμματα μπορούμε να στηρίξουμε. Πάντως, ακόμη και στο Αζερμπαϊτζάν, ακόμη και στη Λευκορωσία, ασχολούμαστε και με θέματα μεταρρυθμίσεων. Στο Αζερβαϊτζάν έχουμε θέματα διαφοροποίησης της οικονομίας. Στη Λευκορωσία κάνουμε τα πρώτα βήματα για να μεταρρυθμιστεί ο επιχειρηματικός κλάδος. Ε, πάντως, ήδη επιχειρούμε κάποιες συστημικές αλλαγές. Και στη Γεωργία και την Ουκρανία έχουμε στηρίξει συνολικές μεταρρυθμιστικές φιλοδοξίες των χωρών αυτών. Και μάλιστα, ενώ ξεκινάμε από το κεκτημένο το ευρωπαϊκό, που σίγουρα δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει άμεσα και περισσότερο όλες τις χώρες, περνάμε λοιπόν από το κεκτημένο περισσότερο σε αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, στην Ουκρανία, αποκέντρωση, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενεργειακός μετασχηματισμός, σημαντικές αλλαγές. Περνάμε λοιπόν από τα προγράμματα στη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και της, μεταρρύθμι... της μεταμόρφωσης, του μετασχηματισμού της χώρας. Δεύτερον, ε, ενισχύουμε τη σχέση μας με την κοινωνία των πολιτών, με τα think tank, με τους παρόχους υπηρεσιών. Αναβαθμίζουμε αυτές τις σχέσεις και στηρίζουμε τους παράγοντες, τους φορείς μεταρρύθμισης στις χώρες αυτές με επαναπροσανατολισμό των κανόνων μας ε, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο που μπορούμε να στηρίζουμε όχι μόνο τους συνήθεις υπόπτους, αλλά ε, να φέρουμε την ενίσχυση και εκτός των πρωτεύουσών στις ε, ΜΚΟ, στην κοινωνία των πολιτών, σε τοπικούς φορείς και παράγοντες. Τρίτο, με ε, τον πρώην και τον είναι επίτροπο, επενδύουμε και οικονομικά. Προσπαθούμε ε, και τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνούς ε, χρηματοπιστωτικούς φορείς να τους φέρουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Και συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς για να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές τις χώρες από κοινού. Αυτές είναι πολύ σημαντικές αλλαγές λοιπόν της πολιτικής μας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση. Και οι προτεραιότητες της ΡΙΓΑ και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2020 που περιμένουμε στους τέσσερις ε, άξονες, στις τέσσερις βασικές κατηγορίες, ε, είναι διαφορετικά πια. Και στην περίπτωση της Ουκρανίας κάναμε και ένα βήμα επιπλέον, γιατί έχουμε και την ομάδα στήριξης για την Ουκρανία, που είναι ένας μοναδικός φορέας και είναι η μοναδική ομάδα εργασίας που έχει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια χώρα εκτός των συνόρων της, εκτός της επικράτειάς της. Και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ομάδα στήριξη για την Ουκρανία, για να πειραματιστούμε σε όλα αυτά τα θέματα και δεχομένω να τα εφαρμόσουμε και σε άλλες χώρες. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για τις συμφωνίες που αρχικά εκπορευόταν από το κεκτημένο και που δεν ενδιαφέρεται τόσο, δεν ενδιαφέρε τόσο τις χώρες αυτές γιατί είχαν άλλες ανάγκες. Ξεπεράσαμε όμως αυτό το στάδιο του κεκτημένου και το αντισταθμίσαμε με μεγαλύτερη συμμετοχή στις μεταρρυθμίσεις. Αυτά και ίσως πιο διεξοδικά αργότερα στη συζήτηση. Να σας δώσω και κάποια παραδείγματα για το τι κάναμε με τη νέα προσέγγιση. Ένα παράδειγμα που ανέφερε συχνά ο πρώην Επίτροπος είναι ότι σε μία περιοχή του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου που έχει μεγάλες συναλλαγματικές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το, στηρίξαμε τις, τις μισές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό νόμισμα στηρίζοντας τους εταίρους. Άλλο παράδειγμα, όπως πολύ εύστοχα είπε και η Αντζελίνα, θα πρέπει να δούμε και τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η νέα πράσινη συμφωνία είναι κάτι που ήδη εφαρμόζαμε ενεργά με τεράστιες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, μαζικές επενδύσεις στις τοπικές υποδομές, ε, διαχείριση αποβλήτων, λιμάτων, καθαρό νερό, επενδύοντας στις αστικές συγκοινωνίες, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Κάτι που δεν κάναμε πριν από 3-4 χρόνια. Οπότε έχουμε πρόοδο και θα λάβουμε υπόψη και τις προτεραιότητες της νέας γεωπολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, για το μέλλον. Γι' αυτά που λέει και η Αγγελίνα, υπάρχει ένας πολύ δραστήριο σε δημόσιους διάλογους ε, και υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο πλαίσιο που αναδύεται την επόμενη δεκαετία, το οποίο αφορά την ανθεκτικότητα. Μία έννοια που μπορεί πραγματικά να είναι πολύ ωφέλιμη για όλα τα σκέλη των σχεδίων μας. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ενέργεια, Για την ε, Ουκρανία, λοιπόν, αν είχαμε πρότυπα ενεργειακής απόδοσης ε, στα επίπεδα της ευρωπαϊκής χώρας που έχει τις ε, χαμηλότερες επιδόσεις, και δεν θα αναφέρω εδώ συγκεκριμένα, τότε δεν θα χρειαζόταν να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όλο αυτό, λοιπόν, συνδέεται και με άλλες πτυχές. Κοινωνική αντοχή και ανθεκτικότητα είναι πράγματα στα οποία θα πρέπει να επενδύσουμε. Φυσικά, διακυβέρνηση, κράτος δικαίου, να συνεχίσουμε τις πιέσεις ε, για την ε, περαιτέρω εκδημοκράτηση της χώρας. Όλα αυτά μας αφορούν και θα μας απασχολήσουν. Κλείνοντας, πολλά λέγονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, διαφοροποίηση, εναντί της ε, συμπερίληψης. Εμείς από την Επιτροπή τα εξετάζουμε πιο πρακτικά τα πράγματα. Έχουμε δύο πλαίσια. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι το περιφερειακό πλαίσιο ενός ευρύτερου εγχειρήματος ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που αφορά και την Ανατολή, αφορά και τον Νότο, έχει και περιφερειακή διάσταση και διμερή. Στη δεμερή διάσταση και πάλι έχουμε ε, σε μεγάλο βαθμό διαφοροποίηση μεταξύ χωρών. Εμείς λοιπόν από πρακτική άποψης δεν βλέπουμε πρόβλημα να έχουμε και ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο και για τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, το οποίο όμως δεν μας εμποδίζει καθόλου να κάνουμε και αυτή τη διαφοροποίηση που συνήθως σε πρακτικό επίπεδο προκύπτει από τις διμερείς σχέσεις με τις χώρες. Και εκεί μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Θα μείνω εδώ ή μάλλον δύο πράγματα ακόμα. Εκτιμούμε ιδιαίτερος ε, τη στήριξη του Κοινοβουλίου και μελών του, πολλά από τα μέλη της ΑΦΕΤ αλλά και ευρύτερα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστηρίζουν ο φίλος μας, ο κύριος Κουμπίλιους, δημιούργησε και το φόρουμ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και μας βοηθάει και στην στρατηγική μας επικοινωνία. Το το ορισμένοι, εδώ χωλαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα είχαμε τον Brexit αν ήμασταν καλύτεροι στην επικοινωνία. Έχουμε επενδύσει πολλά σε αυτή την προσπάθεια. Να δώσουμε ένα όνομα ε, στην συνδρομή που παρέχουμε με το λεγόμενο EU4 Energy, EU4 και συμπληρώνουμε τον τομέα πολιτικής. Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν επικοινωνούμε ε, σε ένα ουδέτερο πολιτικά πλαίσιο. Ε, υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση, ιδίω σε αυτή την ε, περιοχή του κόσμου. Ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ε, γνώμες, πληροφορίες, παρατηρήσεις, προτάσεις για το μέλλον από τις ε, πρωτεύουσε ε, των ε, ανατολικών μας εταίρων, από την πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Ινστιτούτα Ανάλυσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε με πολλά και ενδιαφέροντα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Πρώτος μεταξύ ίσων βεβαίως Κάλεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους ε, προσκεκλημένους μας. Σημερίζομαι την πλειονότητα των όσων ε, υπόθηκαν. Το σημαντικό είναι όλα αυτά βέβαια να τα διαβιβάσουμε και πέραν αυτής της αίθουσας. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και αυτές οι χώρες έχουν αλλάξει πολύ την τελευταία δεκαετία. Εν ώψη και αυτής της συνόδου, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, αποτέλεσμα που δεν θα είναι φιλόδοξο και ότι θα έχουμε απλώς μία επανάληψη των όσων είχαμε πριν από 10 χρόνια. Δεν γίνεται. Αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία μας. Μετά πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε με σωστά βήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες αυτών των χωρών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακολουθήσει τη μέθοδο Μονέ για πολλά χρόνια. Ε, κάνουμε το, επόμενο βήμα όταν χρειαστεί. Όμως, ε, εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι ακολουθούμε μια τέτοια προσαρμοσμένη ε, μέθοδο. Πρέπει όμως να πείσουμε και τις 27 χώρες να πάρουν ομοφόνος μια απόφαση να ανοίξουμε και τις δυνατότητες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, ιδίω ό,τι αφορά την ομοφωνία. Όμως με αυτά τα συμπεριληπτικά και ολοκληρωμένα προγράμματα, γιατί δεν πρόκειται για επιμέρους και μεμονωμένα έργα, αλλά για ολοκληρωμένα προγράμματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές χώρες είτε προχωρούν είτε έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν ταχύτερα και να μας προσεγγίσουν πιο γρήγορα. Αυτό λέω σε αυτές τις χώρες. Το καθεστώς της υποψηφιότητα δεν πρόκειται να σας φέρει αυτομάτως ε, πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε και την Τουρκία τι έγινε με την Τουρκία, ήρθαν πιο κοντά ή απομακρύνθηκαν, παρότι ήταν και υποψήφια χώρα. Τι έγινε και με την ε, Μακεδονία ε, και το 2005, παρότι άλλαξε τώρα και το όνομά της ε, Βόρεια Μακεδονία. Δεν πρέπει λοιπόν αυτές οι χώρες να μένουν μόνο ε, στην επίσημη ονομασία και στο επίσημο καθεστώς, αλλά στην ουσία, στο πόσο μας προσεγγίζουν. Επομένω, θα πρέπει εκ των πραγμάτων αυτές οι χώρες ε, να έρθουν πιο κοντά προς εμάς, να αυξήσουμε την αλληλεξάρτηση σε ό,τι αφορά τις ε, υποδομές, να γίνουν λοιπόν ε, απαραίτητοι εταίροι σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγμή ε, τι να κάνουμε φυσικά και θα πρέπει να τους αποδεχθούμε. Αυτά μέσω και μακροπρόθεσμα. Ας μείνουμε σε όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα που αναφέρθηκαν. Η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντικό να εμπλακεί Όλα αυτά εντάσσεται στην προσπάθεια για την αύξηση της ανθεκτικότητας. Και όπως είπε η κυρία Σάρη, και μου άρεσε, πρέπει να επικαιροποιήσουμε αυτούς τους νοητικούς χάρτες για την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστούμε. Δεν τους έχουμε προσφέρει τη δυνατότητα να ενταχθούν και να γίνουν μέλη, αλλά καλώς αναφέρατε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις εισηγήσει σας. Πολύτιμες. Να κοιτάξουμε λίγο το μέλλον. Νομίζω μια καλή λέξη είναι η αντοχή, η ανθεκτικότητα. Αλλά αν δούμε τα θέματα αντοχής, θα πρέπει να δούμε και την ψυχολογική ανθεκτικότητα των χωρών αυτών, τη δυνατότητα αντίστασης. Βασική μου ανησυχία είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την κινητοποίηση των πολιτών, ε, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά των ίδιων των πολιτών στις χώρες αυτές για να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, για να έχουν τη διάθεση να προχωρήσουν σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όμως ο κόσμος δεν πείθεται έτσι εύκολα. Βλέπουν και τις εμπειρίες τους από το παρελθόν, από τις γειτονικές χώρες. Γι' αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ με τον κύριο Βοτσοκόφσκι. Αποφεύγουμε για γεωπολιτικούς λόγους να μιλήσουμε για τη δυνατότητα ένταξης. Αλλά αυτό είναι μια επιπλέον πρόκληση. Πώ να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ στην ψυχολογική του δυνατότητα αντίσταση, να προχωρήσουν στι μεταρρυθμίσει. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τι πολύ επιτυχημένε εμπειρίε μα από την κεντρική ας πούμε, Ευρώπη. Η δυνατότητα της ένταξης ήταν αυτό που κράταγε τη δική μας δυνατότητα αντίστασης και την επιμονή μας σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είχαμε μια σαφή προοπτική, μια ξεκάθαρη προοπτική της ένταξης. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα. Και ένα δεύτερο. Εάν δει κανεί την ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων 30 ετών. Έχουμε τα παραδείγματα της κεντρικής Ευρώπης, μια δεύτερη σειρά παραδειγμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά. Για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, νομίζω αυτά τα παραδείγματα είναι θετικά. Είναι χώρε της Ανατολικής Γειτονίας που πρέπει να αναφέρονται πιο συχνά. Να τους δίνουμε το παράδειγμα των Δυτικών Βαλκανίων, να κοιτάμε πώς μπορούμε το παράδειγμα αυτό να το μεταφέρουμε στην Ανατολική Γειτονία. Και πρέπει να βλέπουμε και τι αντιδράσει στην πράξη. Αν αρχίσουμε να κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό, το τι έγινε στα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί και να εφαρμοστεί στι χώρε τη Ανατολική Γειτονία. Τότε ίσω να αποδεχθούν καλύτερα αυτά που του ζητούμε και να προχωρήσουν. Η δική μου λοιπόν επιθυμία είναι να ασχοληθούμε πάρα πολύ με την ψυχολογική ε, αντίσταση και ανθεκτικότητα των χωρών αυτών. Δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμόσει τι μεταρρυθμίσει. Ο κόσμο αισθάνεται μια κόποση εάν δεν βλέπει γρήγορα τα αποτελέσματα. Και εάν δεν τους δείξουμε κάποιον ε, μεγάλο, λαχταριστό στόχο, σαν καρότο, δεν θα θέλουν να προχωρήσουν. Πρέπει λοιπόν και ο υπατός εκπρόσωπος να τα σκεφτεί όλα αυτά. Και κάτι άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η μεθοδολογία της διεύρυνσης. Μια προϋπόθεση μια προϋπόθεση που είχε θέσει και για τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο η Προεδρία του Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει και λίγο ο τρόπος με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Ο κύριος Μαριανή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τους έξι προσκεκλημένους μας και αυτό που είπε η κυρία Σαρή είναι ότι εδώ και 10 χρόνια έχει αλλάξει το όλο σκηνικό, η όλη νοοτροπία. Υπάρχουν νέοι παράγοντε. Βλέπουμε πόσο δραστήρια είναι η Κίνα στη Λευκορωσία. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και όταν λέω ότι υπάρχουν νέοι παράγοντε, ε, εξεπλάγει. Που δεν άκουσα να μιλάει κανείς για την Ευρωσιατική Οικονομική Ένωση στι ομιλίε σα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια οικονομική συνεργασία που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρία από τα έξι κράτη τη Ανατολική Γειτονία συμμετέχουν. Η Λευκορωσία, η Αρμηνία είναι μέλη, η, η Μολδαβία είναι συνδεδεμένη. Η Ρωσία είναι σαφώς ένας εταίρος που πρέπει να έχουμε υπόψη. Αλλά το ερώτημα που θέλω εγώ να κάνω για να περάσουμε από ένα αστείο σε ένα άλλο. Άκουσα κάποιον από τους ομιλητές να μιλά για κράτη ομήρους της Ρωσίας. Μήπως προσπαθούμε να τους κάνουμε ομήρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μήπως τελικά μια τρίτη επιλογή είναι να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, την ιδιαίτερη ιστορία και παράδοση των χωρών αυτών και τους ιδιαίτερους πληθυσμούς που έχουν ε, αυτή είναι η τρίτη ίσω εναλλακτική. Ακούω τον συνάδελφο να λέει ότι θα πρέπει να του δώσουμε την προοπτική τη ένταξη και ίσω αυτό να επιτρέψει να προχωρήσουμε. Όμω το αίτημα των πληθυσμών αυτών είναι διαφορετικό. Ζητούν πρώτα απ' όλα την οικονομική ευημερία, ζητούν ασφάλεια, ζητούν να του ακούμε. Κάποιε φορέ λοιπόν παθιαζόμαστε και μα πιάνει ενθουσιασμό αμέσω με κάτι μικρά δείγματα. Η πρώτη σύνοδο ε, ε, στο ημικύκλιο στην οποία παρέστην ήταν για να ακούσει την κυρία Σαντού. Όμως, εγώ ήμουν από τους λίγους ομιλητέ τότε που έλεγα ότι θα κρατήσει έξι μήνες η όλη προσπάθεια για την Μολδαβία. Ε, όσοι γνώριζαν την ε, κατάσταση στη Μολδαβία ήξεραν ότι είναι δύο φατρίε αυτές που συνεργάζονται και μια τρίτη τελικά έλαβε και την εξουσία. Ε, το ευρωπαϊκό όνειρο, όταν είχα έρθει στο εμεκύκλο και είχε γίνει αυτή η παρουσίαση για τη Μολδαβία, φάνταζε ένα μακρινό όραμα. Ε, μην ξεχνάμε λοιπόν τι θα πρέπει να γίνει με την Ευρωσυντική Οικονομική Ένωση. Αυτό να το λάβουμε υπόψη και κανεί δεν μίλησε για την ομιλία του κυρίου Αλιέφ 23 Δεκεμβρίου, νομίζω, στην τηλεόραση τη χώρα του. Τι είπε σήμερα, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπα που κυκλοφορεί σε αυτές τις χώρες. Αυτό που είπε για τη χώρα του λοιπόν ε, ήταν χρειάζεται το Αζερβαϊτζάν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Χρειάζεται Ευρωπαϊκή Προπτική, Όχι. Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες όπω υπόθηκε για τις χώρες αυτές. Αυτές που έχουν πολύ στένε σχέσεις με τη Ρωσία γιατί είναι εμπλεγμένες ε, Λευκορωσία, Μολδαβία και Αρμενία. Και η Ουκρανία είναι η μόνη από τι χώρε που επέλεξε να ε, έρθει τόσο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιπε ψάχνουν το δρόμο του. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι το εξή. Δεν θεωρείτε ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, να έχουμε ασφάλεια, οικονομική ευημερία, χωρί να είμαστε απαραίτητα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω χρειάζεται να βρούμε την τρίτη οδό. Την τρίτη οδό που θα πρέπει να είναι ραμμένη και κομμένη στα ε, μέτρα και τι ανάγκε των χωρών αυτών. Για να παραφορμή από τα λόγια τη προηγούμενη ομιλητή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δική του ιστορία, την πραγματικότητα των πληθυσμών εκεί και όχι τι δικέ μα επιθυμίε. Και ένα συμπέρασμα, γιατί κάποτε ήμουν και πρόεδρο τη Γαλλική Βολή ε, στην ομάδα Γαλλία-Ουκρανία. Ε, τότε που ο κ. Ζαχόφ ήταν πρωθυπουργό τη Ουκρανία, τι μου είχε πει. Μου είχε πει πάμε ε, στον τοίχο, πάμε σε εμφύλιο πόλεμο. Διότι από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει συμφωνία και απόσταση από τι συμφωνίε που έχουμε με τη Ρωσία και καλύτερα θα ήταν να έχουμε μια ε, στενή εταιρική σχέση ε, με δύο συνεργάτε, όχι με έναν. Ε, εάν συνεχιζόταν αυτό έλεγε θα πάμε σε εμφύλιο πόλεμο. Βλέπουμε τώρα τα σφάλματα του παρελθόντο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια στους εμπειρογνώμονες που μας παρουσίασαν την κατάσταση της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Με μεγάλο επαγγελματισμό από ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την πραγματική εικόνα της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες που έφυγαν από την ε, Σοβιετική Ένωση και για τη τελική ανάλυση η ανατολική εταιρική σχέση τους δίνει την ευκαιρία να διαλέξουν αν θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Μόσχας ή θα προτιμήσουν τη δυτική λύση, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποσχέσεις ε, που δώσαν προς χώρες αυτές ήταν πάρα πολλές και ευρύτατες και το βασικό στοιχείο είναι ότι η ανατολική εταιρική σχέση τους δίνει και από πολιτική άποψη τη δυνατότητα να παίζουν στο ένα ή στο άλλο γήπεδο, στο ένα ή στο άλλο ταμπλό. Και σίγουρα μια εταιρική σχέση με τρεις ε, εταίρους δεν θα λειτουργήσει στο μέλλον. Οι πολιτικοί θα επιδιώξουν την α για να μείνουν σε μια τελωνιακή ένωση της Ρωσίας ή αργά ή γρήγορα να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι κατά ανάγκη το γεγονός ότι οι Μολδαβοί, οι Ουκρανοί δεν ξέρουν τι θέλουν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν τους δίνουμε μία ξεκάθαρη λύση και προοπτική για το μέλλον. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Μολδαβοί, ο λαός της Μολδαβίας για παράδειγμα, τα έχει λίγο χαμένα με τα κόμματα. Γιατί θέλουν κάποια κόμματα να είναι στην Τελωνιακή Ένωση της Ρωσίας, ενώ η Μάγια Σάντου είναι πιο φιλοευρωπαία και θέλει τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κανένας δεν τους θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Μόσχα από τη μια λέει δεν έχουμε σύνορα και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν είναι ώρα τώρα να συζητούμε για διεύρυνση και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που μπορεί να είναι αλήθεια γιατί ε, γύρω μας έχουμε τα ευρασιακά στρατεύματα. Το θέμα είναι όμως να δώσουμε μια προπτική μελλοντική στις χώρες αυτές. Η Μολδαβία θα γίνει μια μέρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέω για αύριο, έστω μετά από 50 χρόνια αλλά έστω μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη προοπτική στη Μολδαβία για το μέλλον. Η δεμή το παιχνίδι μεταξύ Μόσχας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρυξελών θα συνεχίσει να κρατά τη χώρα σε μια αβέβαιη κατάσταση. <coughs> σε μια μετέωρη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιορτάνοφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Русия оказва влияние върху политиката на страните от източното партньорство. Η Ρωσία ασκεί τεράστια επιρροή στις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Και το κάνει αυτό με προπαγάνδα και με διαφθορά των πολιτικών ελίτ. Είναι αναφίβολο ότι η, διαφορά, η διαφθορά στις χώρες αυτές φέρει τη σφραγίδα της Ρωσίας. Οι οικονομικές ελίτ των χωρών αυτών έχουν περισσότερες σχέσεις με τη Ρωσία παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία παρέχει όπλα και οργανώνει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Έτσι ενισχύει την επιρροή της και προωθεί τα συμφέροντά της η Ρωσία στην περιοχή. Γι' αυτό ε, έχουν χάσει και τον μπούσουλα οι πολίτες των χωρών και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πέραν των οικονομικών ε, δυσχεριών που υφίστανται, έχουν και την προπαγάνδα να τους ταλανίζει. Και μάλιστα την προπαγάνδα τη δέχονται και από τους ντόπιου πολιτικούς. Ένα μεγάλο, ένας μεγάλος αριθμός των πολιτικών των χωρών αυτών εξυπηρετούν τα προσωπικά τους ιδιωτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του λαού τους. Και ξέρουν ότι τα προσωπικά τους συμφέροντα θα προωθήσουν μόνο μέσω της Μόσχας. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ανήμπορες και προσκρούν στα συμφέροντα των πολιτικών και στην εξουσία του χρήματος. Βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο λοιπόν. Τι θα, τι θα κάνουμε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δίλημα αυτό δεν πρόκειται να το λύσει να το λύσουν προγράμματα ή διαδικασίες. Το δίλημα αυτό μπορεί να λυθεί, να μόνο χάρη σε μια καινοτόμη προσέγγιση και σε ενατοριστικές πολιτικές σε καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι προς τις χώρες αυτές και να πούμε απερίφραστα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον οι χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα ολοκληρώσουν την πορεία τους και θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στις χώρες αυτές. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε κυρίως τις χώρες που ήδη έχουν αναγγείλει τις ε, ευρωπαϊκές τους προθέσεις και τον φιλοευρωπαϊκό τους προσανατολισμό, όπως είναι η Ουκρανία και η Μολδαβία. Η Ρωσία, βέβαια, θα ενοχληθεί από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να εντάξουμε την κοινωνία των πολιτών στη συζητήση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλο συνάδελφο το λόγο, οπότε θα ζητήσω από το πάνελ, από τους εμπειρογνώμονές μας, μέσα σε ένα δίλεπτο καθένας, να απαντήσουν αν το επιθυμούν. Ποιος θα είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, ο κύριος Γερασίμτσουκ και για τις παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ευγνωμοσύνη μου, κυρίως προς τους κυρίους Κομπίλιος, Μπασέσκου και Γιορτάνοφ, γιατί και οι τρεις στάχθηκαν υπέρ της ενταξιακής προοπτικής των χωρών αυτών, που είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν έχουμε ακόμη τη συνένεση όλων των χωρών μελών υπέρ ε, της ένταξης. Το θέμα είναι Μπορεί να συνδυαστεί η ένταξη ως περιφερει... στην περιφερειακή πρωτοβουλία και στην περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε καταρχήν την πρωτοβουλία των τριών και στην ε, διάσκεψη κορυφής του Βουκορεστίου ήταν ε, σαφής η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την πρωτοβουλία αυτή και σίγουρα οι χώρε Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καθεστώς παρατηρητή σε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, είχαμε την πρωτοβουλία Βουκουρέστι 9, που επίσης ανοίγει τις θύρες στις χώρες ανατολικής γειτονίας για να αποκτήσουν τουλάχιστον καθεστώς παρατηρητή. Και έχουμε το V4, V4 ΣΥΝΕ διαδικασία και συνεργασία με τις χώρες του Βίσεγκρα, ε, τις του Βίσεγκρα είναι σημαντική. Ε, και επαναλαμβάνω στην Ουκρανία δεν έχουμε εμφυλίο πόλεμο. Είχαμε την επίθεση της Ρωσίας, την εισβολή της Ρωσίας. Θα πρέπει να το τονίσουμε. Δεν ήταν εμφύλιος ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Χάρηκα που ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε μαζί μας σε ορισμένα ζητήματα. Η συμμετοχή είναι σημαντική, ως μέλος δηλαδή, η ένταξη. Είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να έχει και την πρωτοκαθεδρία. Κάτι που έχω κατανοήσει τα τελευταία χρόνια, σε αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από ιστορική άποψη, ε, αποτελεί αποτέλεσμα μιας ε, διακρατικής συνεργασίας. Και φυσικά υπάρχει ε, το οικονομικό σκεπτικό όλης αυτής της συνεργασίας, να διευκολύνεται δηλαδή η συνεργασία ε, διασυνοριακά. Όμω, εάν υπάρχει αυτή η συνεργασία, ιδίω με τι χώρες τη ανατολική Εταιρική σχέση, χωρί να τις διαβρύνουμε στις υπηρεσίες, στο εμπόριο, δεν έχει πια νόημα. Όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο οικονομικός χώρος βάσει και της βαλκανικής εμπειρίας. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δεν ισχύουν από μόνοι τους. Λειτουργούν στην πράξη μόνο αν υπάρχει αλληλεπίδραση, ε, αν υπάρχουν συναλλαγές, ανταλλαγή σε εμπορικό επίπεδο, σε υπηρεσίες και το καθεξής. Και είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε ε, πολιτικές, διπλωματικές και τεχνικές ε, δυνατότητες. Δεν έχουμε μόνο την έλλειψη δυνατοτήτων σε διοικητικό επίπεδο. Πολύ συχνά η διαφθορά είναι αυτή που εμποδίζει αυτές τις χώρες. Επομένω, πρέπει να εργαζόμαστε και σε πολιτικό, τεχνικό και διπλωματικό επίπεδο. Πρέπει να εμπλέξουμε λοιπόν τους αρμόδιους ε, φορείς και εμπειρογνώμονες. Και μετά χρειαζόμαστε και καλύτερα θεσμικά όργανα για την διαχείριση της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Euronest, κοινά ε, θεσμικά όργανα εταιρική σχέση πρέπει να εξυγχρονιστούν και να αποτελέσουν ένα καλύτερο βελτιωμένο πλαίσιο. Ο κ. Κακάτσια. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, επί της διαδικασίας εξευρωπαϊσμού. Είναι μία μακρόπνοη διαδικασία. Κατανοούμε ότι δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη Ταυτόχρονα, κάποιος έθεσε υπάρχουν και άλλοι τρόποι πέραν της ένταξης. Η ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης μας έχει δείξει ότι η διεύρυνση ήταν το πλέον επιτυχημένο μοντέλο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα κατανοούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γεωπολιτικές ε, ε αντιπαλότητες μεταξύ Ρωσίας και άλλων χωρών. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να εμπλακεί σε όλο αυτό. Όμως, εάν σταθούμε μόνο στα ευρωπαϊκά συμφέροντα εδώ, οι Ρώσοι δημιουργούν τέτοια προβλήματα ε, σκοπίμως, όπως στην Ουκρανία. Γιατί ξέρουν ότι αν δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα, θα δημιουργήσουν προσκόμματα στην ε, διαδικασία ένταξης αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε πιο ρεαλιστικά την ε, δυνατότητα ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αλλά αυτό ισχύει και για τη Ρωσία. Ξέρουν ότι δημιουργώντα προβλήματα ε, παρεμποδίζουν τη διαδικασία διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα υπάρξει και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, μερικέ παρατηρήσει. Φυσικά και δεν υπάρχει σήμερα εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, χάρη και στι κοινέ προσπάθειε που έχουμε κάνει σε αυτή τη χώρα, έχουμε ε, καταφέρει να αποφύγουμε τις ε, συγκρούσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορες αντιθέσεις βέβαια σε πολλά επίπεδα, αλλά είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί και πρέπει να το θυμίζουμε και μεταξύ μας και μεταξύ των πολιτών. Ποια είναι η δική μας συμβολή δηλαδή στην αποτροπή του πολέμου και στην οικοδόμηση της ειρήνης. Ναι, είναι καλή ιδέα να ε, επενδύσουμε περισσότερο στην προσέγγιση Ζαμονέ, όπω είπε και ο κύριο Γκάλερ προηγουμένω. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε και στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ένα καλό ε, μηχανισμό για να δράσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Κύριε Κομπίλιο, ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις σας προηγουμένως για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα όσα κάνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια και στις ε, χώρες της Ανατολικής Εταιρικής ε, Σχέσης. Μιλήσατε για τη δικασία του Βερολίνου, τη γνωρίζω καλά. Το θετικό και η χρησιμότητά τους είναι ότι κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά με τους εταίρους, με ε, τον EEA, τους εξωτερικούς εταίρους, μια μεγάλη διεύθυνση και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην ε, Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και δύο λόγια για την ε, μεθοδολογία διεύρυνσης. Ο υπότος εκπρόσωπος ε, θα τα παρουσιάσει όλα αυτά στις αρχές Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά αυτή τη στιγμή με πολύ θετικό τρόπο και είναι σημαντικό. Πρέπει πάντα να βλέπουμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερως ε, τις επόμενες εβδομάδες, εμάς και στη συνέχεια και εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πολύ σημαντική η συμβολή σας. Για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, η Αρμενία ολοκλήρωσε μία ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ε, ήταν και μέλος ε, της Ευρασιατικής. Δεν ζητούμε από τους εταίρους να επιλέξουν ή εμάς ή τους άλλους. Για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά εδώ στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, κατά τη γνώμη μας, να σεβαστούμε απολύτως τις επιλογές ε, των εταίρων. Αρκεί, αυτό λέμε εμείς μόνο, όσα κάνουν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να συμμορφώνονται με τους ε, κανόνες μας, τη νομοθεσία μας, το διεθνές δίκαιο και το καθεξής. Αυτό ακριβώς λέμε και στις συζητήσεις μας. Ξεκαθαρίζουμε και πάλι, δεν απαιτούμε από τους ε, εταίρους να διαλέξουν ανάμεσα σε εμάς και άλλους εταίρους. Μπορούμε να εργαστούμε σε πολλά επίπεδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις, γιατί η Αντζελίνα αναφέρθηκε στη μεθοδολογία της διεύρυνσης, που θα παρουσιαστεί και τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αφορά αυτό που ανέφερα προηγουμένω στη Συμφωνία σύνδεση. Η μεθοδολογία που στηρίζεται στο κεκτημένο. Το κεκτημένο όμω δεν φέρνει τις μεταρρυθμίσει που χρειάζονται οι χώρε η τι αλλαγέ που στηρίζεται στο πολίτε. είναι το πρόβλημα. Και αυτό που θέλουμε και στα Δυτικά Βαλκάνια είναι τα θεμελιώδη πρώτα. Μεταρρύθμιση των θεσμών, τη δικαστική εξουσία, της ε, ε, οικονομική κατάσταση, επανασυμφιλίωση μερικέ φορέ όπω στα Βαλκάνια. Θα γίνει μια προσπάθεια λοιπόν να κάνει, γίνει μια ανακατάταξη των προτεραιοτήτων και να αναδείξουμε τα θέματα που δεν σχετίζονται με το κεκτημένο. Γιατί το, το ΑΚΙ δεν είναι το σχέδιο στρατηγικής για να καλύψουμε τα ουσιώδη, τα θεμελιώδη ζητήματα και δεν ανταποκρίνεται στις ειδικέ ανάγκες κάθε χώρας. Φάνηκε αυτό και στη Συμφωνία Σύνδεσης και στη ενταξιακή διαδικασία, στη διαδικασία διεύρυνσης. Δεύτερον, και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν γίνεται. Δεν έχουμε εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε την επίθεση, την εισβολή της Ρωσίας και θα πρέπει να είμαστε σαφείς, κατηγορηματικοί και ξεκάθαροι και να το επαναλαμβάνουμε γιατί ακόμη αναφέρεται μερικές φορές η κατάσταση ως εμφύλιος πόλεμο στην Ουκρανία. Και μερικές φορές είμαστε ητοπαθείς στην Ευρώπη, ότι χάσαμε την ε, δύναμη επιρροής μας. Αλλά ακόμη και χωρίς ε, την προοπτική της ένταξης, σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ιδιαίτερως σε πολύ εντυπωσιακέ ε, δημοκρατικές αλλαγές στην Ουκρανία. Και το γεγονός ότι σε μια, χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, ο πρόεδρος που είχε όλες τις εξουσίες ε, της ιδιότητάς του δεν έκανε τίποτα για να κερδίσει εκλογές ε, ε, και είχαμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας, αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και ε, μεγάλη επιτυχία της Ουκρανίας και αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε γιατί αυτή την επιρροή μας ε, να συντελούμε αλλαγές τη χρησιμοποιούμε ακόμη και χωρίς την υπόσχεση της ένταξης σε καμία περίπτωση βραχυπρόθεσμα άλλωστε και αυτό το γνωρίζει ο κόσμος της περιοχής. Υπάρχουν και κάποια δυσάρεστα ίσως ναι, αλλά υπάρχουν και ευχάριστα και θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να τα επενούμε ιδιαίτερως. Επίσης, κάποιος πρότεινε η εταιρική σχέση να γίνεται μεταξύ τριών μερών. Ε, και αυτό. Ε, αλλά τριγωνικές σχέσεις ε, δεν είναι το κλειδί ισχυρών εταιρικών σχέσεων κατά τη γνώμη μου. Το τρίγωνο πολλές φορές είναι προβληματικό. Και κάποιοι συνάδελφοι που ε, ε, ε, ασχολούνται με τα θέματα αυτά στα κοινωτικά θεσμικά όργανα πολύ πριν από μένα, μου είπαν ότι πρώτα στη Ρωσία προσφέραμε την ανατολική εταιρική σχέση, αλλά απέριψε την πρόταση. Δεν έγινε η ανατολική εταιρική σχέση κατά της Ρωσίας ή βάρος της Ρωσίας. Απλώς η Ρωσία δεν είχε συμφέρον για κάτι τέτοιο και διαφόρησε. Και στη συνδιάσκεψη του Μονάχου άλλαξε πορεία. Ε, και επαναλαμβάνω, όπως είπε και η Αντζελίνα, δεν προσφέραμε την ε, ανατολική εταιρική σχέση ε, κατά της Ρωσίας, της βάρος της Ρωσίας. Πρώτα την προσφέραμε στη Ρωσία, άλλωστε. Ευχαριστώ. Και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της συζήτησης, του χρόνου της συζήτησης, ίσως έτσι τελευταία στιγμή να είχαμε κάποια τελικά συμπεράσματα από τον κύριο Πέτρας Αουστρεβίτσιους Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φοβερή συνεισφορά της όλης συζήτηση στην έκθεση του Κοινοβουλίου για την Ανατολική Γειτονία. Ιδέες και πορίσματα στρατηγικής σημασίας. Προτάσεις ιδιαίτερα σημαντικά. Μαζί με τους Κεώδης θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα ενσωματώσουμε στο τελικό σχέδιο τη έκθεσης. Αν δούμε την ανατολική γειτονία μπορούμε να αναγνωρίσουμε ε, κάποια απλά αλλά σημαντικά στοιχεία. Στην ε, περιοχή αυτή έχει περάσει η παγκοσμιοποίηση και έχει εκτεθεί σε διαφορετικούς κινδύνους, πολιτικούς, οικονομικούς, δημερών σχέσεων, λόγω του μεγάλου γείτονα εξανατολών, εξανατολάς, Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αντιστραφεί, δεν είναι δυνατόν να την αποφύγουμε και δεν στρεφόμαστε κατά του ανατολικού μας γείτονα, αλλά υπέρ των ε, γειτόνων μας τα ανατολικά. Να είμαστε όμως και ειλικρινεί. Ό,τι επιτυχία, ό,τι επίτευγμα και αν ε, καταφέρουν οι χώρες της ανατολικής γειτονίας θα έχουν τεράστια επίδραση στο τι θα συμβεί στη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας να τις αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων ας πούμε και με τη Ρωσία. Δεν θέλουμε να απειλήσουμε με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, τη Ρωσία, αλλά να πάρουν μια δημοκρατική κατεύθυνση και όχι την απολυταρχική. Η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία έχουν ήδη περάσει σε μια καλύτερη κατάσταση. Όμως θα πρέπει να προσαρμόσουμε και την εργαλειοθήκη μας, την πολιτική και οικονομική εργαλειοθήκη μας. Χρειάζεται χρήμα για να μετατραπούν σε κάτι δημοκρατικότερο τα καθεστώτα εκεί. Και την θεσμική διοργάνωση. Θα πρέπει εκεί να ποντάρουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας να είναι σταθερά μελλοντικά μέλη, αξιόπιστοι εταίροι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους τους προσκεκλημένους ομιλητές για τις σημερινές τους εισηγήσει και ευχαριστώ και τους ε, εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων που ήρθαν σήμερα για να συνεισφέρουν. Ταυτόχρονα και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Προσβλέπω στην επικοδομητική συνεργασία μας για να συντάξουμε το σχέδιο έκθεσης και να ε, προωθήσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ευχαριστώ κύριε Αστραβίτη, ευχαριστώ όλου του συναδέλφου που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ όσου ήρθαν ω προσκεκλημένοι ομιλητέ για να μα προσφέρουν τη δική του θεώρηση για τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ το μέρο αυτό τη συνεδρίαση λίγη. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, after a hopefully... Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την ενδιαφέρουσα και παραγωγική ακρόαση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βίτολτ ε, Βαστσικόφσκι που προέδρευσε στο πρώτο τμήμα και να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίαση, το σημείο 11 που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Γεωργία ε, και κατά μήκο των διοικητικών συνοριογραμμών και θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό Κέτα Βανσίκη Υπουργό Επανασυμφιλίωσης και ισότητα των Πολιτών και τον κύριο Κάχα Κουτσαβά, Αντιπρόεδρο της ε, Γεωργιανής Βουλής. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους καλεσμένους μας από τη Γεωργία Αντιλαμβάνεστε ότι η Επιτροπή μας παρακολουθεί εκ του σύνεγγης ε, τις εξελίξεις στην πατρίδα σας και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία. Οι δύο καλεσμένοι μας θα μας ενημερώσουν για τις πρόσφατες εξελίξεις μέχρι τις 12 ακριβώς μετά θα αποχωρήσουν, θα μας ενημερώσουν για την προβληματική κατάσταση κατά μήκο και κοντά στις διοικητικές συνοριογραμμές στις υπορωσική κατοχή ε, περιοχές Απχαζίας και Νοτιού Αιτίας. Είχαμε πρόσφατα πολλές ταραχές και είχαμε και τις πρόσφατες εξέλιξεις στην Τυφλίδα, κυρίως ε, το σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Θα δώσω πρώτα το λόγο για 10 λεπτά στην Υπουργό της Γεωργίας και μετά στον Αντιπρόεδρο της Βουλής για 10 λεπτά καθένας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση που με απευθύνετε, καθώ και για το γεγονός ότι μου δίνετε το λόγο σήμερα για την πολύ σημαντική πρόκληση στην Γεωργία με ε, ε, τη συνεχιζόμενη κατοχή των εδαφών τη από την Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν έχουμε μία παγωμένη σύγκρουση, δεν πρόκειται για μία στατική κατάσταση υπάρχει μια αρνητική δυναμική σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Απχασία, η Νότια Οσετία, όλο ένα και περισσότερο απομονώνονται και στρατιωτικοποιούνται. Ο αριθμό ε, των στρατιωτικών δυνάμεων έχουν αυξηθεί σε 10.000, ενώ έχουμε ε, σημαντική απώλεια σε ό,τι αφορά τον ε, τοπικό πληθυσμό. Η πλειονότητα βρίσκεται σε εξορία, δεν έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν, ενώ άλλοι φεύγουν ε, ε, εξαιτία των κακών ε, οικονομικών προοπτικών. Υπάρχουν 130 στρατιωτικέ δοκιμέ κάθε χρόνο σε αυτέ τι περιοχέ. Ιδίω στην Νοτέα βλέπουμε ένα πληθυσμό μόλι 20.000 και ουσιαστικά πρόκειται για μια στρατιωτική βάση και μόνο. Έχουμε πάνω από 100 επωνομαζόμενες συνθήκες που υπογράφονται μεταξύ Μόσχας και των ε, ε, αρχών που υιοθετούν ε, τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, ρωσικό έλεγχο στην περιοχή αυτή ό,τι αφορά τον ενεφοδιασμό. Είχαμε τη συμφωνία ΣΥΦΑ το 2008, 50 γύρι διαπραγματεύσεων στη Γενέβη με παρουσία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των Ηνωμένων Εθνών προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα για την μη χρήση θεωτικής ε, δύναμης ε, από την Ρωσία και την επιστροφή των εκτοπισμένων. Σε ένα εξαιρετικά δυσχερές ε, περιβάλλον, εμείς ε, διατηρούμε την προσήλωσή μας για να διερευνήσουμε δυνατότητες προόδου σε μια συνεχή ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά ζητήματα. Επί ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη αυτής της διαδικασίας που θα είναι κρίσιμη σημασία και για το μέλλον. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αποστολή παρακολούθηση που έχει έναν ειδικό και πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό ρόλο επιτόπου. Συνεχώς ασκούνται πιέσεις ε, για πρόσβαση στις ε, κατεχόμενες περιοχές. Ξέρετε ότι αυτό δεν επιτρέπεται μέχρι τώρα, είναι απαράδεκτο. Και φυσικά και υπάρχουν και κάποιες πολύ λυπηρές ε, ενέργειες κατά των μελών της αντιπροσωπείας. Στις 24 Οκτωβρίου λοιπόν του 2019 η επωνομαζόμενη ΚΑΚΕΜΠΕ της Νότιου Οσετίας ε, προειδοποίησε κατά των ε, ε, περιπολιών στις περιοχές που αλέγχονται από τη Γεωργία. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ ενσχετική κατάσταση συνοριοποίηση στην περιοχή του τελευταίου μήνε. Θέλουν να πάνε πέρα από τη γραμμή των κατεχομένων και να αποκτήσουν τον έλεγχο σημαντικών περιοχών υπό τον κεντρικό κυβερνητικό έλεγχο και μάλιστα ακολουθούν και μία αυστηρή ρητορική ε, όπου εκδίδουν τελεσίγραφα και απαιτούν απόσυρση των, ε, της παρουσίας. Επιπλέον, έχουν, ε, κρατούν ομήρους απλούς πολίτες για να πετύχουν αυτούς τους στόχους τους. Εδώ και πέντε μήνες το μόνο ε, σημείο σύνδεσης ε, της περιοχής με τη Δυτική Γεωργία έχει κλείσει απολύτως. Το Αχαλγόρι έχει 100... 1.500 ε, πολίτες και βρίσκονται πλήρως απομονωμένοι σε μια πλήρη ανθρωπιστική κρίση. Δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, ε, άλλα προϊόντα, στις συντάξεις τους. Ε, έχουμε χάσει ανθρώπινες ζωές για αυτό το λόγο, επειδή δεν τους επιτρέπεται να πάνε στην ελεγχόμενη περιοχή για να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ε, υπάρχουν οικογένειες που έχουν χωριστεί, οι γονείς και τα παιδιά. Η κατάσταση έχει ξεπεράσει ε, κάθε όριο από ανθρωπιστικής άποψης. Δεν μπορούμε να την ανεχτούμε. Εγώ λοιπόν ε, απευθύνω αυτό το μήνυμα προς εσάς να επιτραπεί ε, η επαφή μεταξύ των δύο περιοχών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις. Είμαι πεπισμένη ότι τα μέλη της Επιτροπής σας θα στηρίξουν αυτή την, ε, αυτό το ανθρωπιστικό μήνυμα, να ενώσουμε τις φωνές μας για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την αδικία. Υπάρχουν ε, χιλιάδες ακόμα που πλήττονται από, αυτό τον, από αυτή την απομόνωση. 100 χιλιόμετρα σηματοπλέγματος ε, διαιρούν 116 χωριά στη Γεωργία και καταστρέφουν χιλιάδες ζωές ανθρώπων που ζουν εκεί. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Και χθε το απόγευμα είδαμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να οικοδομούν αυτό το ε, τείχος σε μια περιοχή που ήδη είχε ένα επεισόδιο συνοριοποίησης ε, τον περασμένο Οκτώβριο. Όλα αυτά δημιουργούν επιπρόσθετες ε, προκλήσεις από ανθρωπιστικής άποψης και από πλευράς ε, εδαφικής ακαιρεότητας, ιδίως πέραν του συρματοπλέγματος. Το 2018 και 2019 είχαμε τρομερές συλλήψεις εξαπλάσεις ελλείψεις σε μια προσπάθεια να περάσουν από μια πλευρή στην άλλη. Και πλήττονται όλοι από αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήμουν στις Βρυξέλλες, είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω. Το θέμα ενός ε, πολύ γνωστού γιατρού που συνελήφθη τον Νοέμβριο υπήρξε μεγάλο ε, ενδιαφέρον διεθνώ και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σα γιατί καταφέραμε να επιλύσουμε την, ε, το πρόβλημα αλλά είχαμε εκατοντάδε άλλε τέτοιε ελλείψεις ε, τα τελευταία 8 χρόνια και με τραγικές καταλήξεις σε κάποιες περιπτώσεις. Τέσσερις νεαροί έχασαν τη ζωή τους και οι δράστες ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι. Δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη. Αυτό δείχνει ε, πόσο δεινή είναι η κατάσταση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή φύγεται και πόσο πρέπει ε, να αξιοποιήσουμε και τα διεθνή ε, μέσα. 40.000 άνθρωποι είναι θύματα αυτής της κατάστασης. Ε, πλήττονται από ξεκάθαρη εθνική διάκριση, τα βασικά τους δικαιώματα στην ιδιοκτησία, ε, στην ε, ελεύθερη μετακίνηση, στην εκπαίδευση, στην μητρική τους γλώσσα, όλα αυτά πλήττονται. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το 2014 που ο, ο, ο τέος, πρόεδρος της ε, αναγκάστηκε πλέον να, να παραιτηθεί. Υπήρχε τρομερή δυσαρέσκεια. Η σημερινή κατάσταση λοιπόν δεν ε, ωφελεί κανέναν, ούτε τους ε, Γεωργιανούς, ούτε τους, κατασ... τους κατοίκους της ε, Απχασίας ή της Οσετίας, ούτε καν της Ρωσίας θα έλεγα. Και για τους λόγους που προανέφερα, τα τάγκς και τα σερματοπλέγματα δεν προάγουν μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά μας. Αυτή είναι η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή σήμερα. Ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν είναι δεν τυχαίο ότι όλη αυτή η εταιρική σχέση στην Ανατολή ε, ε, συνδέεται με τις ε, ανεπίλητες συγκρούσεις του παρελθόντος. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη δική μας συμβολή. Αμετάκλητη πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σίγουρα δεν ενεργούμε σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Η διατήρηση της ε, σταθερότητας και της ειρήνης είναι ε, μία μακρόπνοη προσπάθεια. Υπάρχουν τρομερές προκλήσεις, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι κρίσιμη σημασία ε, η συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Το θεμέλιο είναι σταθερότητα, ειρήνη και η επίλυση διαφορών. Διάλογος, συμφιλίωση σε σχέση με τις κοινότητες της Απχασίας και της Οσετίας. Αυτή είναι η βασική πυλώνες. Εμείς έχουμε μια ειρηνευτική πολιτική που ενεργεί προδραστικά. Φυσικά προσπαθούν, η, η άλλη πλευρά προσπαθεί να υποκινήσει τεχνητές ε, προκλήσεις. Όμω θέλουμε να βοηθήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς να προστατεύσουν ε, τα δικαιώματά του, να βελτιώσουν το βιωτικό του επίπεδο, και να δημιουργήσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης παρά τις ε, τεχνητές διαιρέσεις. Ε, δημιουργήσαμε μια νέα πρωτοβουλία λοιπόν, ένα βήμα προς ε, ένα καλύτερο μέλλον που παρέχει διόδους εμπορίου, εκπαίδευσης, περίθαλψης και άλλων πλευρών που άπτονται του περιβάλλοντος, της γεωργίας και το καθεξής χέρι διεθνού στήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερω. Και το Κοινοβούλιο ομόφωνα υποστήριξε αυτό το ε, ειρηνευτικό πλαίσιο και μπορώ να σας πω ότι παρότι βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο και παρά τις ε, δυσκολίες υπάρχουν σαφή δείγματα ε, προσήλωσης και των δύο πλευρών και της Απχασίας και της Οσετίας. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Το 2019 έχουμε 2,5 φορές περισσότερους ε, φοιτητές από την Αυχασία και Οσετία που έχουν πρόσβαση ε, στην ανώτερη εκπαίδευση χάρη σε αυτές τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες. Και με την πρώτη πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος λάβαμε 15 φορές περισσότερες αιτήσει για εκπαιδευτικά προγράμματα. Μιλάμε για εκατοντάδε ε, αιτήσει. Πολύ μεγάλος αριθμός για τόσο μικρές κοινότητες. Τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς ε, όλα αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη. Είναι μια ευκαιρία να επενδύσουμε ε, στην ειρήνη με την κοινωνική επαφή και το διάλογο. Ξεκινήσαμε ένα νέο οικονομικό μηχανισμό, το Ταμείο Ειρήνης, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα εξυπηρετεί αυτούς ε, τους σκοπούς και θα ενισχύει τη συναλλαγή μεταξύ των εταίρων. Ακόμα και με ε, μικρή συνεισφορά μπορούμε να έχουμε μεγάλο αντίκτυπο. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα κεντρικό ρόλο στην ενευτική διαδικασία. Σας είμαστε ευγνώμονες για όλες ε, τις υπάρχουσες δομές ε, συνεισφοράς και φυσικά θέλουμε να διερευνήσουμε και άλλες δυνατότητες ε, υποστήριξης αυτών των νέων ευκαιριών υπό το Γεωργιανό Σχέδιο Ειρήνης. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας λοιπόν για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες σε αυτή την ενευτική διαδικασία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την σταθερότητα και την ειρήνη και στη Γεωργία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Ε, με ευγνωμοσύνη λοιπόν βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τον Ιούνιο του 2018 Δέκα χρόνια μετά τη ε, ρωσική εισβολή αναφέρει ξεκάθαρα ότι η συνεχιζόμενη κατοχή γεωργιανών ε, εκτάσεων είναι ε, κάτι το κατακριτέο και η επίλυση των διαφορών στη Γεωργία είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο συνολικά. Η Γεωργία διατηρεί την προσήλωσή της περισσότερο από ποτέ προς ε, ε, την Ευρωπαϊκή της οδό και αυτό είναι μια ξεκάθαρη δέσμευση της κυβέρνησης και του λαού μας. Το 83% του λαού υποστηρίζει αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Υπερασπιζόμαστε λοιπόν την επιλογή μας για την ελευθερία. Και αυτό εντάσσεται στην, στο θεματολόγιο της Γεωργίας για την πρόοδο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και για την επίλυση διαφορών. Και η αμοιβαιότητα είναι πολύ σημαντική. Εγώ φέρω το παράδειγμα των κοινών επιτευμάτων μας για την ε, άρση των, της υποχρέωσης θεωρήσεων. Δεν έχει να κάνει μόνο με την δυνατότητα των πολιτών μας ε, να ταξιδεύουν χωρίς ε, θεωρήσεις. Είναι και το πολύ σημαντικό μήνυμα και αυτή η ξεκάθαρη αίσθηση των πολιτών μας ότι ανήκουν στην Ευρώπη και έτσι αποτελεί μία ελπίδα και μία φιλοδοξία για ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε μερικά μέτρα παραπέρα, να μιλήσουν με τους γείτονές τους, γιατί υπάρχουν αυτά τα τεχνητά τείχη που πρέπει να καταρριφθούν. Σας ευχαριστώ πολύ και φυσικά είμαι στη διαθεσία σας για ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την εισηγησή σας και τώρα, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για την ευκαιρία να σας απευθυνθώ. Να απευθυνθώ στους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τους φίλους και συνεργάτες μας τα αποτελέσματα της συνάντησης για τις σχέσεις ήταν σημαντικά για την ενισχυμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Ο σκοπός είναι να παραμείνουν οι ανάγκες μας προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα. Την περασμένη, τον περασμένο Σεπτέμβριο αναλάβαμε την Προεδρία της Υπουργικής Συνόδου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μιλάμε για χώρε που θέλουμε να επιστρέψουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό ε, εδώ και δεκαετίε. Τώρα όχι απλώ είμαστε ένα από τα πιο επιτυχημένα κράτη στην ευρωπαϊκή αυτή πορεία, αλλά καταφέραμε να έχουμε μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή κοινότητα. Δεν θα μιλήσω για τις απειλές από την Ρωσία, υπόθηκαν ήδη πολλά γι' αυτό. Απλώς να πω ότι τα προηγούμενα 200 χρόνια η Ρωσία είναι υπαρξιακή πραγματικής ε, ε, υφής απειλή στην ε, Ρωσία. Κατέχει το 20% του εδάφους μας και έχει παραβιάσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες. Υπονομεύει όχι μόνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά είναι μια απειλή ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή. Η διαρκής υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας είναι ουσιαστική για την καταπολέμηση και την πάυση των, το διχασμό αυτό. Η Ευρωατλαντική Συμμαχία επίσης υποστηρίχθηκε με δημοψήφισμα την πλειοψηφία του λαού. Και το θέμα είναι να γίνει ε, σεβαστεί η βούληση του λαού της Γεωργίας, όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με πρακτικά βήματα. Έχουμε ε, έρθει πιο κοντά από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύνδεση συμφωνίας και την ε, σφαιρική και ενισχυμένη συμφωνία συνεργασίας. Είμαστε στατηγικοί εταίροι. Έχουμε ξεπεράσει το 34% ως προς την απελεύθερωση της κυκλοφορίας και ένα δις Γεωργιανοί έχουν από τη στιγμή εφαρμογή του συστήματος ταξιδέψει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συμμετοχή στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, σχετικούς οργανισμούς και φορείς και η συνεργασία μας είναι πραγματικά πολύ στενή. Η εξωτερική πολιτική της Γεωργίας. Οι ευρωατλαντικές μας προσδοκίες έχουν πλέον γίνει επίσημες με την ανάλογη συνταγματική αλλαγή ε, για το Σύνταγμα τώρα στη Βουλή μας Έχουμε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας για να ξεκινήσει μια πλήρη συνταγματική μεταρρύθμιση και να υπάρξει σύγκληση του συνταγματός μας με τις βασικές αρχές του Διεθνούς ε, Συνταγματικού Δικαίου να προσαρμοστεί το συνταγματικό μας σύστημα στα μακροπρόθεσμα δημοκρατικά ε, συμφέροντα. Η μεταρρύθμιση ε, ολοκληρώνει την τελική μετάβαση της γεωργίας στην κλασική κοινοβουλευτική δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου. Βασιστήκαμε στις εξής αρχές. Κοινοβουλευτισμός, ισχυρό κοινοβούλιο, αποτελεσματική κυβέρνηση και ανεξάρτητος δικαστικός κλάδος. Η ειδική ε, συνταγματολόγοι για την μεταρρύθμιση τόνισαν την ανάγκη εκπόνησης νέων ιστορικών κανονισμών για να υπάρξουν επιπλέον εχέγγυα για την ε, ε, λογοδοσία του Κοινοβουλίου και την διαφάνεια. Δηλαδή η εκτελεστική εξουσία να μπορεί να λογοδοτεί. το 2019 ήταν εξαιρετική χρονιά γιατί είχαμε δραματική αύξηση τη λογοδοσία τη εκτελεστική εξουσία με προσωπικέ μαρτυρίε και ε, συνομιλίε και ενώπιον επιτροπών του Κοινοβουλίου. Το 2018 έγιναν συνταγματικέ αλλαγέ και είχαν ήδη εγκριθεί προκειμένου να υπάρξει ένα μεικτό εκλογικό σύστημα με μεικτή αναλογική που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2024. Οι αλλαγέ βασίζονται στην Ειδική Επιτροπή του ΑΣΕ για την ε, Ερηνή Σύνοδο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πολιτική συμφωνία για όλα τα θέματα αυτά ήταν ευρεία και η εκλογική μεταρρύθμιση ήταν επιτυχής παρά τι παραφωνίε των τελευταίων τριών μηνών. Όπως ξέρετε, προς απογοήτευσή μα, το Κοινοβούλιο της Γεωργίας δεν πέρασε τον νόμο για την αλλαγή κατοχής ε, δεδομένων ε, για τον κλικό νόμο το 2020 με πολύ μικρή διαφορά. Οι προτινόμενε αρχές της πρωτοβουλία φάνηκαν να μην είναι αποδεκτές για ένα μεγάλο μέρο των βουλευτών για το σύστημα διακυβέρνηση με την πλειοψηφία ε, που είχε προταθεί και να πω ότι είχαμε τη δυνατότητα δύο φορές στο παρελθόν να περάσουμε στο σύστημα της απλής αναλογικής ως Γεωργία ε, και θα το είχαμε ήδη το 2020 έτοιμο το 2014, το 2017 και δυστυχώ δεν είχαμε αρκετή υποστήριξη, αρκετέ ε, ψήφου από άλλα κόμματα. Και ακόμη και αλλαγέ που προτίθηκαν το 2018 όταν τελικά προτάθηκε ξανά το σύστημα έπλης αναλογική, δεν υποστηρίχθηκε από καμία, με καμία ψήφο από κανένα άλλο κόμμα. Το τωρινό σύνταγμα που προώθησε το κόμμα Georgian Dream, το όνειρο τη Γεωργίας, θέλει να φέρει τη μεταρρύθμιση ει πέρασμα το 2024, με το σύστημα να είναι πλήρως θεμητό. Το κόμμα μας είναι δεσμευμένο να φροντίσει να υπάρξουν ανεξάρτητε, αμερόληπτε και δίκαιες εκλογές στο 2014. 2024. Οι συνταγματικέ αλλαγέ το 2019 προκάλεσαν αντιδράσει από την αντιπολίτευση και του υποστηρικτέ του. Μάλιστα, κλήθηκαν αυτοί οι υποστηρικτέ και ψηφοφόροι να ε, παρακολύσουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου μπλοκάροντας τι εξόδου και τι εισόδου. Στι γύρω δρόμου υπήρχαν διαδηλώσει. Και την ασφάλεια των διαδηλωτών έπρεπε να αγγιηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, οι διαδηλωτέ μπόρεσαν να οργανώσουν πορεία μπροστά στο Κοινοβούλιο, χωρί όμω να μπλοκάρουν και να φράξουν τι εισόδου. Ε, είμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε διάλογο, προτείνοντα τα κόμματα τη αντιπολίτευση να περάσουμε σε κοινοβουλευτική μορφή για τη διοργάνωση των συνομιλιών μα και με τη συμμετοχή ε, εκπροσώπων τη κοινωνία των πολιτών και των πολιτικών κομμάτων βάσει των συστάσεων του ΑΣΕ για την ε, εκλογική μεταρρύθμιση. Είμαστε ευγνώμονε στου διεθνεί συνεργάτε μα και φίλου μα για τις προσπάθειες να παρεμβληθούν ως διαμεσολαβητές σε αυτές τις συνομιλίες. Μπορέσαμε με το κυβερνών κόμμα και τους εκπροσώπους αντιπολίτευσης να διοργανώσουμε ε, την εκλογική διαδικασία για το 2020. Ο διάλογος βρίσκεται όμως σε εξέλιξη. Είμαστε πεπισμένοι ότι η σταθεροποίηση της δημόσιας σφαίρας ε, με τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών του 2020 βάσει ελεύθερων δημοκρατικών προτύπων και με ένα ε, σύστημα πλήρους αναλογικής μέχρι το 2024 είναι απαραίτητα να ενισχύσουμε ε, το αμετάκλητο τη διαδικασία μια οικοδόμηση ε, κοινοβουλευτική ανεξάρτητη δημοκρατία στη Γεωργία. Δυστυχώ, η τάση των διαδηλώσεων που διοργανώνει η αντιπολίτευση διωγγώνεται και οδηγείται σε βία επεισόδια. Ε, και τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν σε παραβατική συμπεριφορά την, ε, τους οι διαδηλωτέ ε, κλήθηκαν να ε, εισβάλλουν στο κτίριο της Βουλής. Εκατοντάδε. παρά τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ε, εισέβαλαν στο κτίριο της αστυνομίας απέναντι από το κοινοβούλιο και πέταξαν διάφορα οχήματα παρά την παρουσία των αστυνομικών. 30 τουλάχιστον φύλασαν το κτίριο με ειδικά μέσα, με κράνη και ασπίδες και ε, παρά τι ε, τις καταγγελίες για κατάχρηση βίας από τις διοκτικές δυνάμεις, τρεις αστυνομικοί προσήχθησαν. Υπήρξε πειθαρχική ε, δίωξη, 19 πολιτικοί υποτίθεται κρατούμενοι βάσει των όσων λέει αντιπολίτευση επίσης προσήχθησαν, γιατί προετοίμαζαν βομβιστικές επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια. Και 18 συμμετείχαν σε δύο επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση και οι διαδηλωτέ του έχουν, λέει, δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Οι αστυνομικοί όμω έκαναν χρήση εσωρόπη βία. Δεν υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων των δραστών βάσει όσων γίνονται προς στιγμή. Βάσει των περασμένων γεγονότων, θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή σα στο εξή γεγονό. Όσο και αν εκτιμούμε τη στατική μα συνεργασία και τους φίλου μα, πρέπει να είστε ειλικρινεί μαζί μα και θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενική πληροφόρηση χωρί να δέχεστε την προπαγάνδα ε, των όσων παρουσιάζουν τα γεγονότα διαφορετικά η κοινοβουλευτική σύνοδο Euronest θα πρέπει να δεχτεί το έτοιμά μα στο τελικό τη ψήφισμα να συμπεριλάβει ένα, ψήφισμα, ένα κείμενο για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Γεωργία. Και οι αποφάσει σας θα πρέπει να παραμείνουν βασισμένε σε σαφή αποδεκτικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε που παραμένετε ε, σταθεροί σε αυτή την προσέγγιση για το 2019 επίσης και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος από το Κοινοβούλιο. Η μεταρρύθμιση χαρακτήκε με βάση τις συστάσεις και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, της διεθνούς κοινότητας και των πολιτικών κομμάτων με βασική έμφαση στη βελτίωση του μηχανισμού πλαισίου για την λογοδοσία των δικαστών, το πρωτογενέ δίκαιο, την ε, μεταρρύθμιση τη δικαστική σχολή και το καθεξής. Η δικαστική μεταρρύθμιση ε, έγινε πρόσδεκτη από την Επιτροπή της Βενετίας, ε, την Πρεσβεία της, των ΗΠΑ και των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκής Ένωση μετά από δύο χρόνια έμονων και αδικαιολόγητων επιθέσεων κατά του δικαστικού σώματο και των δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να γίνουν αναξιόπιστοι και να πληγεί η ανεξαρτησία του γεωργιανού δικαστικού συστήματο. Είχαμε και μια πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που δεν βρήκε παραβιάσεις στην εκδίκαση υποθέσεων και το δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Ε, τελικά στην υπόθεση αυτή το πόρισμα του δικαστηρίου έγινε δεκτό και οι κατηγορίες ε, κατέστησαν κενές νοήματος. Όμως βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η κατηγορία ήταν αδικαιολόγητη και δεν μπόρεσε να αποδειχθεί από τους αντιδίκους. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν η υπόθεση δεν έχει οδηγήσει σε... δεν έχει δείξει κάποιο σαφές δείγμα. Ε, θα προσπαθήσω να συντομεύσω, ναι. Να πω και δύο λόγια για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Γεωργία. Τα πράγματα δεν ήταν ποτέ όπως σήμερα. Χρειάζονται δέκα μέρες για να πάρει κανείς μια άδεια και να ανοίξει σταθμό. Μετά το 2012, 7 χρόνια μετά μάλλον, όταν είχαμε μόνο τέσσερις τηλεοπτικούς σταθμούς, τώρα έχουμε 100. 20 από τους οποίους είναι ψηφιακοί ε, σταθμοί. Βάσει του ε, Ελευθερία του Δικτύου 2019 είμαστε μεταξύ των 10 πρώτων χωρών στην Ελευθερία του Διαδικτύου. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διαθεσή μου, οπότε θα πω απλώ τι άλλε μεταρρυθμίσει θέλουμε να διοργανώσουμε στο μέλλον για το κράτο δικαίου και τι έχει πετύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασική προτεραιότητα για την ατζέντα των προτεραιοτήτων στη Γεωργία. 41, ε, είμαστε ε, στον κατάλογο των ε, χωρών Θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης την ε, προστασία ανθρωπίνων, των προσωπικών δεδομένων με τον, ανάλογο λειτουργό, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης, την ολοκληρωμένη νομοθετική ε, ε, μεταρρύθμιση με αποπολιτικοποίηση της αστυνομίας, την αντιμετώπιση υποθέσεων βίας κατά των γυναικών, της σεξουαλικής βίας, τα εγκλήματα κατά των ανηλίκων και τα δικαιώματα των παιδιών. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα ε, προωθήσουμε. Ο κατάλογο των προτεραιοτήτων μα και των τελευταίων μεταρρυθμίσεων έχει αλλάξει πολύ το πρόσωπο τη Γεωργία. Χαιρόμαστε λοιπόν για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει και παραμένουμε δεσμευμένοι στην πορεία του εκδημοκρατισμού. Η ανεξαρτησία τη Γεωργία και η αποκατάσταση τη εδαφική τη ακαιρεότητα είναι προτεραιότητα τη εξωτερική πολιτική τη χώρα για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή μα πορεία και το κυβερνητικό σχέδιο παραμένουμε ε, δυνατοί. Παρακαλούμε στηρίξτε την πορεία μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και πάλι σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τις εντατικές προσπάθειες υποστήριξης της χώρας μου. Thank you, Thank... Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Βουλής. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε και την ενημέρωση για την κατάσταση στη Λιβύη ως ονούπο και ο κ. Πιλώνη είναι περιορισμένο στο χρόνο. 10-12 λεπτά μας έμειναν για τη συζήτηση. Ζήτησαν το λόγο οι Γκάλερ, Καλνιέτε, Γιουκνιεβιτσένη και Λεγκόροβα. Yes, of course, no problem. I can... Κανένα πρόβλημα. Θα διαβάσω μόνο τα ονόματα των ομιλητών που δήλωσαν. Ooh, yes, okay. okay. Uh, Μίξερ Καμπίλιος, Κομπίλιο, Μπάνιον. We start, of course, with Marina Kal Ξεκινάμε με την Μαρίνα Κάλιουραντ, που είναι και πρόεδρος ε, της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ε, με τον Νότιο Κάφκασο. Παρακαλώ, χρόνου φίδου. Προσπαθώ να τετραγωνίσω τον κύκλο με τόσο λίγο χρόνο που έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίζω και τους ε, συναδέλφους από τη Γεωργία στη συζήτηση. Θα κάνω λίγα σχόλια γιατί είμαι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με τον Νότιο Κάφκασο. Θα περιοριστώ στο σημερινό αντικείμενο της συζήτησης, ανταλλαγή απόψεων για τη γεωργία και κατά μήκο ε, των διοικητικών συνοριογραμμών. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πιο διεξοδικά αυτά τα θέματα στην συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί στις 12 και 13 Φεβρουαρίου και ελπίζω ότι η Υπουργό Τικελασφίλη θα είναι παρούσα και στη συνεδρίαση εκείνη. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώ, ε, διαπιστώνουμε ότι οι προκλήσει των ρωσικών αρχών και των αντιπροσώπων του συνεχίζονται στη Γεωργία. Παρά την ε, επίσημη επαναφορά της Ρωσίας στις δομέ του Συμβουλίου τη Ευρώπης. Και μάλιστα μήπω έτσι ξεγελαστήκαμε, μήπω ε, έτσι αφήνουμε τη Ρωσία να συνεχίσει το, την καταστροφική τη πορεία συνεχίζει να παραβιάζει τις υποχρεώσεις ε, ε, της ε, συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός του 2008, συνεχίζει στρατηγικές ασχήσεις, προπαγάνδα, στρατηγική προσάρτηση και διαδικασία συνοριοποίησης. Όλα αυτά συνιστούν τεράστια απειλή για το σύνολο της περιοχής του Νοτιοκαυκάσου, όπως είπαν και οι συνάδελφοι από τη Γεωργία. Οι νέε εντάσει και ιδιαίτερα στη Νέα ήταν πρόσχημα για, την, ε, για το αυθαίρετο κλείσιμο των σημείων διέλευσης και το διχασμό κοινοτήτων που παλιά συνυπήρχαν αρμονικά. Και μάλιστα τον Οκτώβριο του 2019 είχαμε ψηφίσουμε για την απαράδεκτη εμ, σύλληψη ε, αμάχων μελών της Αποστολής Επιτήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται και στα δύο κατεχόμενα, και τη Απχαζία και τη Νεοτίου Οσετία. Και δυστυχώ άνθρωποι χάνουν τη ζωή του γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στο διοικητικό έδαφο τη τυφλίδα ε, και να λάβουν την δέουσα ιατρική περίθαλψη. Και μάλιστα ο θάνατο ε, του δόκτωρα Καπριντασβίλη προκάλεσε τη διεθνή προσοχή. Αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε και τις ε, δεκάδες άμαχων απλών πολιτών ε, των χωριών που αυθαίρετα συλλαμβάνονται και χρειάζεται να πληρώσουν πρόστιμα επειδή περνάν τα κατεχόμενα προς την Γεωργία. Και παρά τις διαμαρτυρίες της διεθνούς κοινότητας, μετά από εντάσεις με την αντιπολίτευση ε, παρετήθηκε ο πρόεδρος ε, της ε, Απχαζίας, χωρίς ευτυχώς χρήση βίας. Αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ασταθής ε, στην περιοχή και θα πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, περιμένοντας την διεξαγωγή νέων εκλογών. Και θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση, να δράξουμε κάθε ευκαιρία και να εκφράσουμε την απερίφραστή μας δέσμευση υπέρ της κυριαρχίας της Γεωργίας και της εδαφικής της ακεραιότητας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και την πολιτική της μη αναγνώρισης των καθεστώτων μαριονετών που δημιούργησε το Κρεμλίνο. Επίσης, θέλουμε μια ειρηνευτική επίλυση των συγκρούσεων, χάρη στη διαπραγμάτευση και τη δημοκρατία και μέσω των διεθνών ε, διαπραγματεύσεων στη Γενέβη και θα ήθελα να λάβουμε υπόψη τους πληθυσμούς και από τις δύο πλευρές των σύνορων, όπως φαίνεται από την ειρηνευτική πρωτοβουλία για ρεαλιστικά βήματα για ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την δήλωσή σας. Είστε επικεφαλής αντιπροσωπείας, σε παραλαμβάνω, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Νότιο Κάφκασο και σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή. Δύο λεπτά τώρα το πολύ στους επόμενους ομιλητές. Ξεκινάμε από τη Σάντρα Καλνιέτε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η Μαρίνα Κάλιοραντ. Εγώ θα σας μιλήσω για την εσωτερική κατάσταση στη Γεωργία, για την πολιτική κρίση που λαμβάνει η χώρα στη Γεωργία. Κύρια κύριε Υπουργέ, είπατε ότι ο κόσμος διαδηλώνει στους δρόμους ε, με υποδάβληση της αντιπολίτευσης. Είχα μακρά πείρα από τα λαϊκά κινήματα και γνωρίζω ότι καμία πολιτική οργάνωση, κανένα κόμμα δεν μπορεί να παροτρύνει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων να κατεβούν στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν. Υπάρχουν πολύ πιο βαθύτερες αιτίε. Είπατε ότι οι Γεωργιανοί στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στην ίδια όμως δημοσκόπηση διαπιστώνουμε ότι ο λαός της Γεωργίας θεωρεί ότι η δημοκρατία έχει παλινδρομήσει στη χώρα αυτή. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ένθερμοι υποστηρικτές της Γεωργίας και είμαστε και αρκετά συγκαταβατικοί απέναντι στην πατρίδα σας. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τη Γεωργία όσο μπορούσαμε, όσο παίρνω από το χέρι μας. Αν όμως συγκρίνουμε την Ουκρανία που έχει, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και παρόλα αυτά χρησιμοποιεί τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενώ εσείς χωρίς να έχετε πόλεμο δεν καταφέρατε να τηρήσετε την υπόσχεσή σας να υιοθετήσετε ένα ε, εκλογικό νόμο της αναλογικής, αυτό δεν ε, είναι επιχείρημα υπέρ της δημοκρατικότητας της γεωργίας. Επίσης, ε, ο Ιβανισφίλη, ο πρόεδρος ε, του ναι. κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, λέει ότι πολλοί ε, ηγέτες αντιπολίτευσης ε, θα περάσουν το χρόνο τους στη φυλακή στο μέλλον. Αυτό το σχόλιο είναι παράδεκτο από ε, τον αρχηγό κόμματος, τον Ιβανισβίλη. Και ο πρόεδρος Μποκερία μετά από μία πενταετή σιωπή έχει και πάλι δίνει να βιώνει η ποινική υπόθεση εις βάρος του. Αυτό είναι νομίζω συμβολικό και δεικτικό της κατάστασης στην Κροατία. Ο Σβέν Μίξερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα κατεχόμενα της Απχαζίας και Νοτιού Οσετίας, συμφωνώ απόλυτα με την Μαρίνα Κάλιοραντ. Πολύ ανησυχητική η τάση που ισχύει ε, ριζοσπαστικοποίηση, ε, ε, συνοριοποίηση, στέρηση των πολιτών από πρόσβαση σε φάρμακα, τροφή, απαγόρευση να χρησιμοποιούν την μητρική τους, απαγόρευση διέλευσης στα εδάφη που τον έλεγχο της γεωργίας. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία και φαίνεται ότι περνάμε σε ένα νέο κύκλο εντάσσεων. Σε ό,τι αφορά την εγχώρια κατάσταση, η κυβέρνηση και το κυβερνόν κόμμα ε, θέσπισαν τις ε, θεσμικές αλλαγές ε, και το νέο σύστημα της αναλογικής από το 2024. Βέβαια, αρχικά είχε μετατοπιστεί επί το νωρίτερο αυτή η προθεσμία και ζητήθηκε να επισπευστεί η εφαρμογή της αναλογικής. Πάντως, ε, είναι αξιέπαινο ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τυφλίδα προσπάθησε να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ του κυβέρναντος κόμματος και της αντιπολίτευσης προκειμένου να διευθετηθεί το διέξοδο, το πολιτικό διέξοδο που υπήρχε. Υπάρχουν και συνταγματικές πτυχές αλλά και ε, νομικές πτυχές. Πού πιστεύετε θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβαστική λύση γιατί ο συμβασμός θα πρέπει να έχει σίγουρα και πολιτική πτυχή. Πώς πιστεύετε ότι θα, θα υπερκεραστεί αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, γιατί υπάρχει μεγάλη πόλωση του πολιτικού σκηνικού που μας λυπεί στην Κροατία, αλλά δεν είναι και ίδιο της Κροατίας μόνο, της, ε, στη Γεωργία, αλλά δεν είναι ίδιο της Γεωργίας μόνο, φέρεται και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε ότι έχουμε μια, μια παταγώδη αποτυχία σε τη αφορά τη διάδοση ε, και την ενημέρωση του κόσμου για την κατάσταση εκεί. Εγώ είχα πάει εκεί στα σηματοπλέγματα και μιλούσα με έναν διερμηνέα, μέσονος διερμηνέα, με έναν αγρότη που είχε χάσει την ε, γη του. Δεν μπορούσε να πάει στα χωράφια του και έτσι έχασε την πηγή του εισοδήματός του και την ταυτότητά του αν θέλετε, γιατί του λέγανε οι Ρώσοι ότι εκεί είχε τεθεί το νέο σύνορο και έτσι ήταν σε ρωσική επικράτεια και όχι σε γεωργιανή, παρότι αυτό ήταν γεωργιανός. Επομένω, υπάρχει αποτυχία σε ό,τι αφορά την ε, ενημέρωση και στην Ευρώπη και αλλού. Ο κόσμος δεν έχει απολύτως καμία γνώση της κατάστασης, ότι η Ρωσία δηλαδή συνεχώς ε, μετακινεί τα σύνορα. Από τη μια μέρα στην άλλη αυτός ο άνθρωπος είδε ένα τείχος να υψώνεται και να χάνει πρόσβαση στη γη του. Πρέπει λοιπόν ε, να ενημερωθεί ο κόσμος για αυτήν την κατάσταση. Η Ρωσία ε, ε, τη γλιτώνει σε πολλά από αυτά που κάνει, επειδή ο κόσμος δεν ενημερώνεται. Ευχαριστούμε από τους Πρασίνους, κυρία Γρηγορόβα. Ευχαριστούμε η Υπουργέ Τσακασφίλη για την ενημέρωση. Συγγνώμη για τον τρόπο που προφέρω τα ονόματά σας. Σας ευχαριστώ ακόμα και για την αναφορά στον ε, γιατρό που κάνατε προηγουμένως. Ε, ε, να ρωτήσω πρώτον για τον δόκτωρα Βάγια ποιος πλήρωσε την, για την απελευθέρωσή του, η κυβέρνηση ή μια ΜΚΟ. Μετά υπάρχει μια νέα κατάσταση σε ό,τι αφορά ε, τον, τις ε, διαδικασίες συνοριοποίησης όπου μαρκάρουν δέντρα 240 μέτρα μέσα στα, στην επικράτεια της Γεωργίας και δεν αφήνουν δημοσιογράφους ή ακτιβιστές να μπουν. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να ενημερώνει τους πολίτες για την κατάσταση. Το κύριο Κουτσάβα, ένα σχόλιο, παύλα ερώτηση. Ελπίζω να είστε εξετάσετε αντικειμενικά ε, την ε, γνώμη μου, γιατί και εγώ έχω πάει εκεί, έχω μιλήσει με κόσμο εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν μπλοκάρουν ε, το κοινοβούλιο με το τείχος της τυφλίδας, αλλά ένα σχόλιο ήταν αυτό μόνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείτε ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι θα συμφωνούσαν μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους υπουργού για την ενημέρωση. Συμφωνώ απολύτως ε, με την ε, δήλωσή σας. Η κατάσταση επιδεινώνεται, όλο ένα και περισσότερο. Εμείς ε, την παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζουμε την κατάσταση. Και για μα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις αποστολέ παρακολούθησης. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε παρά τις ε, πιέσεις ε, της ρωσικής πλευράς και άλλων. Δυστυχώς, θεωρώ ότι η κοινωνία επαγρυπνεί και κατανοεί την κατάσταση όπως την αναφέρεται. Αλλά η ρωσική ιδεολογία κατάφερε να παρισφρήσει στο ε, Γεωργιανό Κοινοβούλιο. Και αυτό οδήγησε σε ένα γύρο ε, διαμαρτυριών. όσο περισσότεροι κρατούμενοι υπάρχουν, τόσο πιο επιθετική γίνεται και η Ρωσία. Ε, εσείς τι προσπάθειες αποκλιμάκωσης θα κάνετε. Καλό θα ήταν να λάβουμε και τα στατιστικά για τον αριθμό των ε, κρατουμένων μετά τις ε, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Ευχαριστώ. Τέσσερις συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στους γεωργιανούς συναδέλφους. 12 και 4 θα λήξει αυτό το θέμα, ό,τι και να γίνει. Επομένω, να είστε σύντομοι για να έχουν χρόνο και οι προσκεκλημένοι μα. Ο κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Μια γρήγορη ερώτηση προ την Υπουργό και πώ φτάσατε στα κατεχόμενα εδάφη για να δώσετε ιατρική περίθαλψη οτιδήποτε χρειάστηκε πέρσι το βασικό θέμα είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος αντιπρόεδρος της Βουλής. Σίγουρα θα υπάρχει πάντοτε υποστήριξη για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Όμως, αυτό πρέπει να συμβαδίζει με το να τηρείτε κι εσείς τις δικές σας πολιτικές υποσχέσεις. Και το να μας παρουσιάζετε την αποτυχία να περάσει η ε, μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην ε, Γεωργία ως επιτυχία του κοινοβουλευτικού συστήματος είναι λίγο υπερβολή. Πολλά πολιτικά κόμματα δεν το θέλαν αυτό. Μήπως λέγατε ε, ουσιαστικά ότι θέλετε να αλλάξει ενώ κρύψατε στα παρασκήνια ότι απέτυχε η μεταρρύθμιση που προτείνατε. Ίσως θα έπρεπε να παραδεχτεί το τι έτσι είναι, αν ε, θέλετε να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή σας πορεία. Ευχαριστούμε κύριο Γκριξμάν. Ευχαριστώ. Βεβαίω έχετε την πλήρη υποστήριξη μας ό,τι αφορά τη ρωσική κατοχή και το γενικό στόχο να κινηθεί η Γεωργία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτησή μου είναι αυτή η περίεργη συγκυρία και την δίωξη μελών της αντιπολίτευσης. Έχετε τον κύριο Μποκέρια, τον κύριο Μένια, πολλούς πολιτικούς ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης που διώκονται ή ανακρίνονται ή ερευνώνται. Η ερώτησή μου λοιπόν έχει να κάνει με τον τύπο, διότι όπως όλοι ξέρουμε η προηγούμενοι ιδιοκτήτε αυτή τη εφημερίδα έχουν χάσει του τίτλου κατοχή σα. Τώρα όμω ο κύριο Γουαράνια, που ήταν ο βασικό ιδιοκτήτη προηγουμένω, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει νέο κανάλι. Και αρχίζει δίωξη εναντίον του, κατευθείαν. Ε, Βεβαίω έχουμε σοβαρού προβληματισμού σε σχέση με την ε, δίωξη κάποιου, μόλι έχει διαφορετικέ πολιτικέ απόψει. Ευχαριστούμε, κυρία Μπλινκεβιτσιένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημαντικό έτο για τη Γεωργία. Θα είναι σαν τεστ του κατά πόσον έχει εκδημοκρατιστεί η χώρα. Βεβαίω, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τι εξελίξει και σίγουρα έχετε πολλού φίλου τη Γεωργία στο Κοινοβούλιο. Όχι από το ένα το άλλο πολιτικό κόμμα, αλλά τη γεωργία. Βεβαίω, θα δούμε κατά πόσο θα περάσετε το τεστ τη δημοκρατία και με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά για μένα ήταν πολύ κακό να ακούω πρόσωπο του κυβερνώντο κόμματο να μιλάει να παραπονείται για την κακή αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στις δημοκρατίες. Οι επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαδηλωτών, αυτά δεν σας βοηθούν, δεν δείχνουν καλή εικόνα της Γεωργίας για να βρείτε και άλλους φίλους στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μπορείτε να βρείτε υποστηρικτές για την ευρωπαϊκή σας πορεία έτσι. Αυτό έπρεπε να πω. Και πραγματικά στέλνω τις σκέψεις μου στους φίλους μου, του and Dream στη Γεωργία και τον κύριο Βανισφίλη. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Δεν θα επαναλάβω όσα υπόθηκαν για την, την εδαφική κυριότητα της χώρας, αλλά για τις επερχόμενες εκλογές. Όταν ε, είχαμε την Σύνοδο Ραν και την Σύνοδο Γιουρονέστ και ήμουν και πρόεδρος εκεί, μιλήσαμε και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήθελα λοιπόν να μεταφέρετε το πολύ απλό μήνυμα στον δικό σας ηγέτη. Ο διάλογος θα φέρει αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα των εκλογών ε, θα είναι καθοριστικά εφόσον υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Χωρίς διαποτελέσματα, αποτελέσματα ε, θα είναι περιορισμένη και η εξοπιστία σας διεθνώς. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν ηγέτες αντιπολίτευση στη Γεωργία που δεν έχουν προσκληθεί στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Για... Σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Ε, δύο λεπτά στον καθένα έχουν απομείνει, γιατί είπαμε δύο και τέταρτο θα ολοκληρώσουμε. Αποφασίστε ποιος θα είναι πρώτος. Δυστυχώ δεν έχω αρκετό χρόνο για να απαντήσω σε όλες τις απορίες. Μερικές ερωτήσεις ε, ε, δείχνουν ότι σε, πολλές, σε μερικές περιπτώσεις ε, υπήρξε παραπληροφόρηση ακόμη και σε εσά. Εγώ δεν ήρθα να σας παρουσιάσω την προσωπική μου γνώμη, αλλά να σας παρουσιάσω και τεκμήρια που συνηγορούν υπέρ αυτών που σα είπα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα. Καταρχήν, για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, και πώς θα προχωρήσουμε στις εκλογές του 2020. Μέχρι τώρα οι προτάσεις ήταν αντισυνταγματικές. Ε, έχουμε δώσει τις αντιπροτάσεις, περιμένουμε τη συνένεση. Και συνένεση σημαίνει ότι και, τα δύο, και δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν. Και για να έχουμε συμβαστική λύση θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις όλες οι πλευρές. Εμείς συμφωνήσαμε και δώσαμε τη δική μας πρόταση που νομίζω ότι είναι καλύτερη δυνατή για τη μεταβατική περίπτωση μέχρι το 2024 που θα έχουμε μια πλήρη αναλογική. Το Γεωργιανό Όνειρο, το κόμμα μας πρότεινε τις συνταγματικές αλλαγές και υποσχεθήκαμε πλήρη αναλογική από το 2024 και μετά. Σε ό,τι αφορά τις δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτών, δεν ισχύει αυτός ο αριθμός, δεν ισχύουν αυτά τα στοιχεία. Και πολλοί νέοι κατέβηκαν στους δρόμους ε, με την πρώτη ευκαιρία όταν είδαν έναν Ρώσο να κάθεται αυθαίρετα ε, στη θέση του Πρόεδρου. Το θυμόμαστε αυτό όλοι. Και αργότερα θέλαμε να σας δώσουμε μια πιο ε, κατάλληλη ενημέρωση όταν οι ηγέτες αντιπολίτευσης προσπάθησαν να αναγκάσουν τους πάντες να επιτεθούν στο κτίριο του Κοινοβουλίου και να παρεμποδίσουν το κοινοβουλευτικό έργο. Αυτά δεν ήταν φημολογίες. Ε, έχουμε αποδείξεις, έχουμε τεκμήρια, ήταν γεγονότα όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο, άκουσα πολλά, αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Είχα πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά ζητήματα να αναφέρω και Είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε περαιτέρω ευκαιρία να συζητήσουμε, να σα παρουσιάσω αποδείξει, αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι δικέ μα απόψει του κόμματό μα. Στηριζόμαστε σε τεκμήρια, σε γεγονότα, σε πραγματικά περιστατικά και όποτε σα βολεύει και έχετε χρόνο, πολύ ευχαρίστω να έρθω για να σα ε, παρουσιάσω διεξοδικά. Πραγματικά έχω μια πολύ, ένα πολύ δύσκολο έργο, Mission Impossible, γιατί έχω ελάχιστο χρόνο και πολλέ ερωτήσει. Συμφωνώ πάντω με τον συνάδελφο ότι Μακάρι να είχαμε την ευκαιρία για να απαντήσουμε διεξοδικά και αναλυτικά σε κάθε ερώτηση, σε κάθε σας παρατήρηση. Μακάρι να μπορούσαμε να σας δώσουμε πιο λεπτομεριακές και αντικειμενικές πληροφορίες για να τις κρίνετε ε, εσείς. Πάντως, ένα γενικό σχόλιο είναι ότι η Γεωργία είναι δεσμευμένη υπέρ της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Γεωργίας είναι προσιλωμένη στη δημοκρατία. Και το περιβάλλον της Γεωργίας είναι δημοκρατικό. Υπάρχει πολυφωνία, ελευθερία έκφρασης, ελεύθερα ΜΜΕ. Όλα αυτά τα εγγυόμαστε στη Γεωργία. Και ό,τι συμβαίνει, είτε είναι της αρισκίας ή όχι κάποιον, γιατί όντω επιδέχεται βελτιώσει το σύστημα, αλλά όλα εντάσσονται στο κράτο δικαίου, γίνονται στα πλαίσια του κράτου δικαίου. Κράτο δικαίου και θεσμική σταθερότητα που επίση ε, έγινε από απέναντι η τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίους μήνες. Οικονομική ανθεκτικότητα και ένα στεναρό πρόγραμμα μεταρρυθμιστικό. Αυτά, αυτές είναι οι πηξίδες της γεωργίας και της, του δρόμου της στην ευρωπαϊκή πορεία. Και είμαστε αμετάκλητη και αμετατόπιστη σε αυτή μας την πορεία. Και φυσικά έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Σας τις είπα και εγώ, γιατί έχουμε καθημερινά προκλήσεις και φυσικά θέλουμε ε, μια ειρηνευτική επίληψη και εμείς δίνουμε τη μάχη μας. Δεν έχει παγώσει αυτή η κατάσταση. Καθημερινά δίνουμε τον αγώνα μας υπέρ της ελευθερίας. Και ελπίζουμε να τον συνεχίσουμε με τη δική σας υποστήριξη, με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για την ανθρωπιστική κατάσταση, για τις ε, καθημερινές ιστορίες των απλών ανθρώπων, των απλών αγροτών που θα πρέπει να γίνουν γνωστές για να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει δεινοπαθήσει από αυτά τα σειρματοπλέγματα που έγιναν ε, το συμβολικό πρόσωπο της ρωσικής εισβολής και κατοχής των τμήματων της γεωργικής επικράτειας από τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας από την ε, Γεωργία. Ελπίζω να περάσετε όμορφα στις Βρυξέλλες. Καλή επιστροφή σας εύχομαι και φυσικά η χώρα σας να ξέρετε ότι θα παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ε, της Επιτροπής μας.